Dear colleagues, I would like to start our meeting. Να ξεκινήσουμε. Δώστε προσοχή. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Θα συνδυάσουμε την παραδοσιακή ακρόαση με την διακοινοβουλευτική συνάντηση. Είναι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο μια ιδιαίτερη συνάντηση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι βασικό μας θέμα είναι ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας, τον οποίο πρέπει να έχουν ή έχουν τα κοινοβούλια. Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο επίπεδο διακυβέρνησης χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η κρίση έχει οδηγήσει σε πολλές μεταρρυθμίσεις που μετέφεραν αρμοδιότητες από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο σε τομείς οι οποίοι παραδοσιακά ανήκαν σε εθνικές αρμοδιότητες ή ήσαν εθνικές αρμοδιότητες. Έτσι λοιπόν έχουμε ιδιαίτερως αυξημένη ευθύνη για τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εποπτεία του εκτελεστικού σώματος από ε, το κοινοβουλευτικά σώματα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα το σύστημα διακυβέρνησης και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και υπάρχουν κοινοβούλια τα οποία δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα στον έλεγχο ο οποίος γίνεται στις κυβερνήσεις τους. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται και η συνάντηση αυτή, έτσι ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι κάνουμε σήμερα και τι θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν τρεις εμπειρογνώμονες με τους οποίους θα ξεκινήσει η συζήτηση για να μας δώσουν τη δική τους προοπτική της πρόκλησης αυτής την οποία έχει να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την εποπτεία του εκτελεστικού. Η διάσταση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σήμερα είναι ο δημοκρατικός έλεγχος. και η δημοκρατία στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Είναι κάτι το καθοριστικό σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα ξεκινήσουμε με την καθηγήτρια Κρίστη Νόιχολτ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ, πολιτικές επιστήμες, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, σχολή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και μετά θα παρουσιάσω και τους υπόλοιπους. Θα ξεκινήσετε κύριε Νόιχολτ, 10 με 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα και ευχαριστώ πολύ και για τα εισαγωγικά σας λόγια. Η μελέτη αυτή ε, συνοδεύεται από μερικές διαφάνειες και βασίζεται στις πληροφορίες που αποκομίσαμε από δύο έργα. Το πρώτο από αυτά μας το ζήτησε η ε, Τσπέντε Κάμερ και η Βουλή των ε, Κατοχωρών. Και το δεύτερο πρόκειται ναι, για μια μελέτη με το όνομα ΟΠΑΙ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω στα επόμενα 10-15 λεπτά είναι να προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα του πλαισίου των πληροφοριών που έχουμε, του πώς έγινε αυτή η μελέτη και να δούμε τα τοπικά μέσα και τις διαδικασίες που έχουμε στη διάθεσή μας και σε εθνικό επίπεδο. Όπως ανέφερε και η Πρόεδρος, υπάρχουν διάφορες ε, διαδικασίες για τα εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε εκείνα να μπορούν να ασκούν έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία και επίσης το τι γίνεται στην πράξη, στην πολιτική διαδικασία, δηλαδή τι γίνεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Βλέπουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια χρησιμοποιούν τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Και θέλαμε λοιπόν να απομονώσουμε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και μετά θα συνεχίσουμε με κάποια συμπερασματικά σχόλια. Περνάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Όπως σας είπα, εδώ βλέπουμε το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Επόμενη διαφάνεια, τα μέσα και οι διαδικασίες που έχουμε. Εδώ πέρα φαίνεται ε, η μεγάλη ποικιλία που υπάρχει. Φυσικά η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως γνωρίζετε, βελτιώνει το δικαίωμα πληροφόρηση ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων από τα θεσμικά όργανα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στα Εθνικά Κοινοβούλια έγγραφα, προτάσει, σχέδια κλπ. Ωστόσο, ο έλεγχο σε εθνικό επίπεδο πάνω στην εκτελεστική εξουσία για τα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι πολύ σημαντικός. Και εδώ η κυβέρνηση παρέχει πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ε, διάφορες ε, τομαϊκές επιτροπές. Ε, μετά κάποια, όχι όλα, τα κοινοβούλια τοποθετούνται μετά ε, τις δηλώσεις των κυβερνήσεών τους στην Κοροπέρι, στο Συμβούλιο των Προτέρων επίσης, εξάντε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να παρακολουθούμε τι γίνεται στο Συμβούλιο. και βλέπουμε ότι έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή, υπάρχει ώρα των ερωτήσεων. Επίσης παρατηρούμε μια τάση εξειδίκευσης μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι υπάρχει η διαδικασία της κίτρινης κάρτας που εστιάζει σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκουμε εξειδίκευση με τη μορφή ειδικών εισηγητών ή ειδικών ε, για ευρωπαϊκά ζητήματα που ασχολούνται με συγκεκριμένα ευρωπαϊκά ζητήματα και ενημερώνουν τις επιτροπές τους. Επίσης, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι υπάρχουν ακόμα βασικές διαφορές ανάμεσα ε, στα κοινοβούλια, στα εθνικά κοινοβούλια, από χώρα σε χώρα ανάλογα με τον έλεγχο που ασκούν στην ε, εκτελεστική εξουσία και στο πότε γίνεται αυτός ο έλεγχος. Ούτε αυτό πρέπει να μας εκπλήσει, διότι από τη συνθήκη της Λισαβόνας και έπειτα το βάρος έχει δοθεί στην, ε, στην ατζέντα, στο θεματολόγιο, στις λευκές ή πράσινες βίβλους. Από την άλλη, πανεπιστημιακή βιβλιογραφία είναι επηρεασμένη και από τον πολιτικό διάλογο και εδώ εμφανίζεται ο όρος mainstreaming, συνεκτίμηση της διάστασης στην ευρωπαϊκή πολιτική, όπου έχει γίνει πιο σημαντικός. Υπάρχουν ειδικέ επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων οι οποίες ασχολούνται με τον έλεγχο σε ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και ειδικέ τομεακές επιτροπές. Μετά, στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά την άμεση ε, ενασχόληση στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Εδώ βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε ορισμένα εθνικά κοινοβούλια να υπάρχουν ε, τομεακές επιτροπές οι οποίες μπορούν να ε, εκδώσουν με ίδια πρωτοβουλία μία αιτιολογημένη γνώμη. Επίσης, ο ρόλος του στην Ολομέλεια είναι επίσης σημαντικό σε αρκετά κοινοβούλια από αυτά που μελετήσαμε και οι αιτιολογημένες γνώμες παίζουν σημαντικό ρόλο. Και αυτό είναι σημαντικό διότι αυτό γίνεται υποπίεση χρόνου δεδομένου μάλιστα ότι δεν επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά επιλογημένες γνώμες στην ε, διαδικασία. Δεν δημιουργούν καθυστερήσεις. Επίσης, παρατηρούμε πως το διοικητικό προσωπικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, η διοικητική υποστήριξη. Επιπλέον, στα πλαίσια του πολιτικού διαλογού, παρατηρούμε ότι οι διαδικασίες είναι λίγο πολύ οι ίδιες ε, στα εθνικά κοινοβούλια. Όμως, ορισμένα συντάγματα περιέχουν τον πολιτικό διάλογο ως ε, αναπόσπαστο μέρος του συντάγματος. Αυστρία, για παράδειγμα. Μετά, βλέπουμε εδώ διαφορετικές πληροφορίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 2010 μέχρι το 2013. Παρατηρούμε μια τάση, έστω και σε αυτήν την περίοδο των τριών ετών, και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι το Σουηδικό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει τις περισσότερες αιτιολογημένες γνώμες και αυτό που παρατηρούμε επίσης είναι ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις ε, αιτιολογημένες γνώμες. Από τη μία διεξάγεται έλεγχο σε όλες τις ε, προτάσεις ή στις περισσότερες από αυτές και από την άλλη την ίδια περίοδο που έγινε αυτό η κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση μειοψηφία. Οι επόμενοι ομιλητέ θα σα δώσουν περισσότερε πληροφορίε για τον όρο των κοινοβουλίων. Εγώ θα περιοριστώ στο να σα πω ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στον αριθμό των ε, αιτιολογημένων ε, γνωμών. Περνάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια όπου θα δούμε την περίπτωση του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας, το οποίο την ίδια περίοδο εξέδωσε τις περισσότερες αιτιολογημένες γνώμες. Και αυτό συνδέεται με αυτά που είπα πιο πριν, με το... η πληροφορία δηλαδή που λαμβάνουμε να είναι ανεξάρτητη, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να πάρει θέση. το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που παρατηρούμε σε αυτήν την διαφάνεια, αλλά και γενικότερα, είναι ότι οι άνοβουλες χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα που τους δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας από τις κάτω Υπάρχουν λοιπόν διαφορές και υπάρχουν και διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους το κάνει κάθε χώρα. Τα μέσα λοιπόν της συνθήκης της Λισαβόνας χρησιμοποιούνται από τις άνοβουλες περισσότερο. Κοιτάζοντας τώρα τις ε, προϋποθέσεις χρήσης του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε κάτι που έχει αναφερθεί συχνά και ε, σε συνομιλίες, σε συνεντεύξεις ε, με πολίτες σχετικά με τον ρόλο που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ορισμένα εθνικά κοινοβούλια δεν θεωρούν πως είναι αρμοδιότητά τους να έχουν άμεση σχέση και διάδραση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης, στην ανάλυση κόστους-όφελους φάνηκε ότι με αυστηρά χρονικά όρια αυξάνεται και η εστίαση σε συγκεκριμένους νευραλγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επίσης βλέπουμε ότι ο μηχανισμός άγκυρης προειδοποίησης εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό του προσωπικού που είναι διαθέσιμο. Τώρα, κοιτάζοντας τον αριθμό του προσωπικού στα κοινοβούλια, βλέπουμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Bundestag, έχει έναν αρκετά καλό αριθμό προσωπικού, επαρκή αριθμό. Και εδώ φυσικά πρέπει να διαρωτηθούμε τι ρόλο ακριβώς έχουν οι κοινοβουλευτικοί υπάλληλοι. Έγιναν κάποιες μελέτες από εμάς και προσπαθήσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις αρμοδιότητες των κοινοβουλευτικών υπαλλήλων. Αυτό που είδαμε είναι ότι στην πλειοψηφία τους είναι σύμβουλοι ή αναλυτές οι διοικητικοί υπάλληλοι παρά διοικητικοί καθ' αυτό. Επίσης βλέπουμε ότι κάποιοι υπάλληλοι έχουν συντονιστικό ρόλο. Επίσης οι σύνδεσμοι είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για την περίπτωση της ενεργοποίησης μιας κίτρινης κάρτας ή της ανταλλαγής πληροφοριών ή ο συντονισμός επίσης. Ο συντονισμός ανάμεσα στα κοινοβούλια έχει γίνει πολύ σημαντικότερος, ιδιαίτερα μάλιστα από τη συνθήκη της Λισαβόνας και έπειτα. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια φαίνονται οι ε, προϋποθέσεις του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Εδώ βρήκαμε ότι ο ρόλος των ε, υπαλλήλων, που, των ελιεζών officers όπως λέγονται, αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, την ομαλή επικοινωνία. Επίσης έχουμε το IPEX, το οποίο είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διάθεσή τους. Ωστόσο υπάρχουν διάφορες ε, απόψεις ότι είναι παροχημένο. Όμως σε γενικές γραμμές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την σωστή χρήση της κίτρινης κάρτας και επίσης υπάρχει και ο συντονισμός και τα λαχή πληροφοριών ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια. Όπως ε, γνωρίζετε η τάση για περισσότερες διακοινοβουλευτικές συναντήσεις έχει επικρατήσει. Καθώς επίσης και η τάση εστίαση σε συγκεκριμένα ε, θέματα όπως το ε, CFSP. Περνάμε τώρα στα συμπεράσματα. αναρωτηθήκαμε στην αρχή εάν το ποτήρι είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο και ποια είναι τα αποτελέσματα της συνθήκης της Λισαβόνας. Βλέπουμε ότι υπάρχει περισσότερη διακοινοβουλευτική συνεργασία, αλλά είναι μόνο μία πλευρά του νομίσματος. Βλέπουμε επίσης περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και Αυξημένε αρμοδιότητε του προσωπικού, του κοινοβουλευτικού προσωπικού. Επίσης βλέπουμε πως ε, η διακοινοβουλευτική συνεργασία μας έχει οδηγήσει σε περισσότερη ε, πολυμορφία. Εάν ένα κοινοβούλιο μπορεί εκτός από τις αρμοδιότητές του να εκδώσει και αιτιολογημένες γνώμες, τις οποίες θα τις συμπληρώσουμε με πρόσθετες πληροφορίες. Θα μπορέσει να ε, ε, ασκεί έλεγχο, να συνοδεύει τον έλεγχο αυτό από πολιτικό διάλογο. Συμπεραίνουμε ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει ένας συνδυασμός όλων των μέσων που έχουν τα κοινοβούλια στη διάθεσή τους παρά η επιλογή ενός. Βλέπουμε επίσης και διαφοροποιήσεις τις οποίες θα αναλύσουν περισσότερο οι επόμενοι ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Νόιχολ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρόζεν, στον κύριο Ολιβιέ Ρόζενμπεργκ από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα κάνω μια γαλλογαλλική παρατήρηση, προσπαθώντας να είμαι αισιόδοξο. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Να το πω κάπως εγώ βλέπω τα πράγματα θετικά. Οι λόγοι για τους οποίους το κάνω αυτό είναι τρεις βασικά. Πρώτον, τα εθνικά κοινοβούλια χρησιμοποιούν τα ελεκτικά τους μέσα Δεύτερον, ελέγχουν όλο και περισσότερο τους πρωθυπουργούς σε ευρωπαϊκά θέματα. Και τρίτον, η έννοια του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. Έγινε μια μελέτη λοιπόν και προσπαθήσαμε να ποσοστοποιήσουμε, έχει κάποια όρια βέβαια αυτό, αλλά προσπαθήσαμε να ποσοστικοποιήσουμε την ευρωπαϊκή δραστηριότητα κατά μέσο όρο για κάθε ένα από τα 40 κοινοβουλευτικά σώματα της Ευρώπης πριν την Κροατία βλέπουμε τη μέση κοινοβουλευτική δραστηριότητα. 45 συνεδριάσεις κατέτος των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σχεδόν μία φορά τη βδομάδα, δουλεύουν δηλαδή, και αυτό σημαίνει ουσιαστικά 68 ώρες, οι γνωμοδοτήσεις των κοινοβουλίων είναι περίπου 35 το χρόνο προς τις κυβερνήσεις και 12 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του βασικού πολιτικού διαλόγου αλλά και στα πλαίσια επίσης του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Σε αυτό συνδέονται οι συζητήσεις στην Ολομέλεια κατά μέσο όρο 13 συζητήσεις ελεγκτικού τύπου πριν από τα αντίστοιχα συμβούλια. Συνεπώς, ακόμα και αν ε, δεν έχουν κερδίσει απόλυτα από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, παρότι υπάρχουν περιορισμοί στην ομοθετική τους δραστηριότητα, προσαρμόστηκαν τα εθνικά κοινοβούλια και ιδιαίτερα μετά από την οικονομική κρίση στα ευρωπαϊκά θέματα, με κάποιες διαφορές βέβαια που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό που με βοηθάει είναι ότι εδώ η πληροφορική δεν σας βοηθάει ε, και θα δείτε πού ε, που βρίσκεται το κάθε ένα από τα κοινοβούλια. Το κοινοβούλιο πάνω δεξιά που έχει τις περισσότερες θεσμικές αρμοδιότητες είναι το της Φιλανδίας. Ανάμεσα στα πολύ δραστήρια κοινοβούλια εθνικά που έχουν ισχυρές εξουσίες είναι η γνωστή ύποπτη Σουηδία, Δανία, Γερμανία, κάτω χώρες, αλλά και χώρες οι οποίες μπήκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Εστονία, η Λιθουανία, Τσεχία. Δεν θα πω ε, τις χώρες που είναι λιγότερο δραστήριες, αλλά παρόλα αυτά οι επιστήμονες ε, θέτουν τον δάκτυλο επί του τύπου των ύλων φυσικά. Βέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα, ε, κάτω σώμα της Σλοβακίας και το Ρουμανικό Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορές ανατολής δύσης, υπάρχει μια βασική διαφορά βορρά-νότου. Γιατί δρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κοινοβούλιο. Καταρχάς, λόγω κοινοβουλευτικής παράδοσης. Δεύτερον, διότι υπάρχει μια κοινή γνώμη, όχι σώνη και καλά ευρωσκεπτικιστική, αλλά που θέλει να δει τι γίνεται στην Ευρώπη. Και επίσης και για λόγους πολιτικής συγκυρίας στην Δανία ας πούμε υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφία και το κοινοβούλιο είναι πολύ δραστήριο. Στην Γερμανία λιγότερο ίσως διότι ή μάλλον και στη Γερμανία είναι δραστήριο διότι υπάρχει κυβέρνηση συνασπισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχα κάνει μια μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια με έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Είχαμε παρατηρήσει και αναλύσει τις δραστηριότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων γύρω από το Συμβούλιο, διότι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση επηρεάζεται όλο και περισσότερο στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η απάντηση είναι θετική, γιατί τα κοινοβούλια είναι δραστήρια την παραμονή του Συμβουλίου ή την επομένη του Συμβουλίου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει σημασία εκλογικά και οικονομικά και αυτό είναι κάτι το οποίο κινητοποιεί τους εθνικούς κοινοβουλευτικούς πέραν κάποιου αριθμού συγκεκριμένου ανθρώπων που ανήκουν στη λέσχη αυτών που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά. Μέχρι τώρα η κινητοποίηση αυτών των κοινοβουλίων δεν έχει οδηγήσει σε μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο. Δεν έχει εμποδίσει ας πούμε να βοηθηθεί η Ελλάδα, δεν έχει εμποδίσει να υπάρξει πιστοτική ένωση, τραπεζική ένωση. Θα δούμε όμως ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης. Βλέπετε ότι τα κοινοβούλια τα οποία είναι δραστήρια σαν φόρουμ συζήτησης είναι στην Ιρλανδία σαν παράδειγμα, τα κοινοβούλια τα οποία είναι δραστήρια σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής, είναι το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Λετωνία και η Σλοβενία και υπάρχουν και κοινοβούλια που δρούν την επομένη εκ των υστέρων. Ε, στα πλαίσια μιας διαδικασίας υπολόγου θα έλεγα, είναι το βρετανικό πρότυπο, άλλα κοινοβούλια σύμφωνα με την γερμανική λογική δρούν εκ των προτέρων, πριν η καγκελάριος ας πούμε πάει στο Συμβούλιο, Λοιπόν, ε, αυτά τα οποία λένε οι πρωθυπουργοί και οι παλιοί πρωθυπουργοί είναι ότι τα ε, εθνικά κοινοβούλια παίζουν ρόλο, ακόμα και στις συζητήσεις τους. Όταν είναι κανένας πρωθυπουργός της Σλοβενία ακόμα και, στην, και κλεισμένων των θερών συνάντηση του Συμβουλίου λέει κοιτάξτε εγώ αυτό δεν το δέχομαι γιατί με εμποδίζει το κοινοβούλιο μου. Τα κοινοβούλια δηλαδή είναι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Τρίτος λόγος για να είμαι αισιόδοξο. Τα εθνικά κοινοβούλια είναι κάτι το σχετικά ε, δύσκολο να προσδιοριστεί σαν παράδοση. Υπάρχουν διαφορετικές κοινοβουλευτικές παραδόσεις στην Ευρώπη. Αρκεί να πάει κανείς στο Westminster, στο Bundestag, στην Assemblée Nationale για να δει ότι ακολουθούνται διαφορετικές παραδόσεις, ε, διαφορετικά μέσα μέτρα και ε, ταυτόχρονα υπάρχουν και πάρα πολλές ομοιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συζητήσεις που προκαλεί στην ουσία δημιουργεί ένα κοινό κορμό συζητήσεων. Η κατηγορία Εθνικά Κοινοβούλια πλέον ε, θα έλεγα έχει εξοικειωθεί με τις συζητήσεις γύρω από τη συνέλευση, γύρω από την αναφορά των κοινοβουλίων στη συνθήκη, από το Μάστριχτ μέχρι τη Λισαβόνα, για την Κοζάκ και για τις στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι αυτή η σχέση είναι δυτή. Από τη μία τα εθνικά κοινοβούλια αντιμετωπίζονται σαν χώροι δημοκρατίας, διότι εκλέγονται άμεσα, διότι συζητούν και διότι είναι πλουαριστικά ε, και οδηγούν σε ε, διαφωνίες, δείχνουν τις διαφωνίες με μεγαλύτερη αν θέλετε ευκολία από ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δύσκολα ξεφεύγει από την ομοφωνία η οποία είναι το βασικό του χαρακτηριστικό η συνένεση μάλλον, όχι η ομοφωνία, η συνένεση. Και υπάρχει μια πολλαπλότητα ρόλων θα έλεγα, που γίνεται αποδεκτή γενικά. Είναι η επόμενη διαφάνεια, πάλι είναι μικρά τα γράμματα, δεν διαβάζονται, αλλά εδώ εξηγούμε τα, πρώτη, τα πρότυπα λειτουργία. Να ελέγχει κανείς το τι κάνει το κοινοβούλιο, αυτό το κάνει ας πούμε η Φιλανδική Βουλή, το policy shaper μορφοποιεί και επηρεάζει τις δημόσιες πολιτικές και στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό ας πούμε το κάνει το γερμανικό κοινοβούλιο. Public forum είναι ένα κοινοβούλιο που γίνονται συζητήσεις, αντιπαραθέσεις. Ε, Ευρωπαίος παίκτη, δηλαδή ένα κοινοβούλιο που θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμα και στην Επιτροπή. Είδαμε τα παραδείγματα της Πορτογαλικής Βουλής και της Σουηδικής Βουλής. Ε, εμπειρογνωμοσύνη κοινοβουλευτική, ένα κοινοβούλιο το οποίο προσπαθεί να είναι ειδικό στα ευρωπαϊκά θέματα. Έχουμε εδώ την Άνω Βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα αυτό ότι κάποια κοινοβούλια δεν επιλέγουν, ας πούμε, το κοινοβούλιο το Σουηδικό παίζει σε όλα τα ταμπλό. Ενώ άλλα κοινοβούλια είναι πρωταγωνιστές σε διάφορους υποτομείς. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες ανάλογα με την πλούσια συνταγματική ιστορία της Ευρώπης, την ιστορία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας εδώ και αιώνες. Πέραν τούτου, και σε μια δεύτερη φάση θα είμαι πιο απεσιόδοξος και θα σας δείξω τις ε, σκιασμένες περιοχές. Ο μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση στον τομέα τη επικουρικότητας. Του ασκώ σκληρή κριτική και δεν είμαι μόνο. Το 90% των ακαδημαϊκών των σχετικών με τα θέματα αυτά είναι εναντίον του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της επικουρικότητας λέγοντας ότι είναι πολύ περίπλοκο, είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ κοινοβουλευτική ενέργεια, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο χωρίς πολύ αποτέλεσμα τελικά είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σε εισαγωγικά εθνικιστικό και δείχνει ένα αρνητικό ρόλο για τα κοινοβούλια ως θεματοφύλακα των εθνικών παραδόσεων. Τα κοινοβούλια θέλουν να λυθούν τα προβλήματα, να αντιμετωπιστεί τρομοκρατία, να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας και να μην μπουν σε διαδικασίες άλλου τύπου. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στις σχέσεις της Βουλής και της Βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με την πρόταση για, ένα κόκκινη, για μια κόκκινη κάρτα η οποία μπορεί να είναι μια πρόταση είτε άχρηστη είτε επικίνδυνη. Στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε τον αριθμό των οδηγιών, των κανονισμών και των αποφάσεων που γίνονται δεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 15 χρόνια. Βλέπετε ότι ήδη το 2010 με την οικονομική κρίση υπάρχει μια τρομερή πτώση και η πτώση αυτή δεν έχει ανακάμψει ακόμα. Το ακούμε αυτό που λένε στο Κοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει πολύ νομοθετική δραστηριότητα στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λοιπόν το Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβραδύνουν την νομοθετική παραγωγή. Ενώ η ίδια η νομοθετική παραγωγή είναι ιδιαίτερα μειωμένη. Λοιπόν, ένα δεύτερος λόγος απεσιοδοξίας και θα είμαι πολύ σύντομο εδώ. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι πάρα πολλά κοινοβούλια στην ουσία εξειδικεύονται ή μάλλον κάποιες μικρές ομάδες, πολύ μικρές ομάδες βουλευτών εξειδικεύονται ε, για τα στα ε, ευρωπαϊκά θέματα. Πολλές φορές μάλιστα οι ίδιοι οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες στην ουσία καπαρώνουν σε εισαγωγικά ε, με τη δράση τους την απουσία της κοινοβουλευτικής, πραγματικής κοινοβουλευτικής δράσης. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Οι εκθέσεις γράφονται, τα ψηφίσματα ψηφίζονται, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή των κοινοβουλευτικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό σε σχέση με το δημοκρατικό ιδεώδες. Η λύση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα είναι το λεγόμενο σύστημα mainstreaming, δηλαδή ένα σύστημα όπου τα ευρωπαϊκά θέματα συζητώνται από το σύνολο των κοινοβουλευτικών επιτροπών και όχι μόνο από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Το Bundestag είναι μια καλή, ένα καλό παράδειγμα. Το δύσκολο είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κινητοποιήσει τους βουλευτές να δραστηριοποιηθούν αν δεν υπάρχει αυτή η εξειδίκευση που τους δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουν διαδικαστικά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, αυτά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι σε σχέση με τις συζητήσεις στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια τα ευρωπαϊκά θέματα στην ουσία κυκλοφορούν περισσότερο και αυτό είναι θετικό. Ένα τελευταίο σημείο απέσιοδοξίας. Η διακυβερνήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύστημα λήψης αποφάσεων έτσι όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την κρίση καθιστά όλο και πιο δύσκολο τον έλεγχο από πλευράς των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τρία παραδείγματα. Πρώτον, οι νομοθετικέ αποφάσει της Ευρωπαϊκή Ένωσης θα πετούν όλο και περισσότερο χρόνο. Έχετε ένα μέσο όρο ε, υιοθέτηση ε, των οδηγιών και των κανονισμών της Ένωσης εδώ και 15 χρόνια. Το 1996 χρειαζόταν ένα χρόνος για να προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία. Πέρυσι χρειάζονταν περίπου δύο χρόνια. Υπάρχει δηλαδή μια ουσιαστική επιβράδυνση της ε, ταχύτητας υιοθέτηση ε, ε, κανονισμών, οδηγιών κτλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τα εθνικά κοινοβούλια γιατί δεν γνωρίζουν σε ποια φάση θα παρέμβουν. Τη στιγμή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τη στιγμή των διαπραγματεύσεων των τελικών. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί δύο χρόνια στην ουσία είναι η μισή διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής θητείας στα εθνικά κοινοβούλια. Κάποια κείμενα τα οποία είναι υποσυζήτηση σήμερα θα γίνουν δεκτά ενώ θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο κοινοβούλιο, μια νέα πλειοψηφία. Δεν υπάρχει δηλαδή συνέχεια από πλευρά τη εξέταση των εθνικών κοινοβουλίων. Ένα άλλο πρόβλημα σε σχέση με την σημερινή διακυβέρνηση της Ένωσης είναι κάποια στοιχεία που γνωρίζετε καλά, ότι δηλαδή οι περισσότερες αποφάσεις στα πλαίσια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας υιοθετούνται στην πρώτη ανάγνωση και όχι στη δεύτερη το 14, το 93, το 93 επαναλαμβάνω τις 100 των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την φάση της πρώτης ανάγνωσης. Αυτό προκαλεί μια δυσκολία για τα εθνικά κοινοβούλια και δεν τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις γιατί είναι μυστικές, γιατί γίνονται στα πλαίσια σκοτεινών τριμερών διαλόγων ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν για τα εθνικά κοινοβούλια και τους ερευνητές, τους δημοσιογράφους, τους πολίτες να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα αυτή. Υπάρχει σε αυτή τη φάση λίγος θεσμοποιημένος πλουραλισμός και αυτό καθιστά την δημοκρατία την κοινοβουλευτική επίσης λιγότερο πλουραλιστική. Συμπερασματικά λοιπόν, φτάνω στο τέλος, στο συμπέρασμα, τέσσερα σημεία μάλλον, Τελικά, τα κοινοβούλια τα εθνικά, όπως σας είπα, είναι δραστήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ περισσότερα από όσο πιστεύαμε και πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Χρησιμοποιούν τις αρμοδιότητες τις οποίες έχουν, στηρίζονται περισσότερο σε σχέση με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και σε σχέση με αυτό το ψευτοσύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Δεύτερον, η επιβεβαίωση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων περνά από τα εθνικά τους πολιτικά συστήματα και από τις δραστηριότητές τους στο εσωτερικό του πολιτικού του συστήματος. Υπάρχουν όμως τρόποι κοινή και συλλογική συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι απόπειρε που γίνονται τώρα σε σχέση με τη λεγόμενη πράσινη κάρτα μου φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικές και νομίζω ότι επιτρέπουν να γίνονται με σταθερή κατά τα άλλα και ε, χωρίς αλλαγές στη συνθήκη. Λοιπόν, στρατηγική τρόμπλογη είναι μια τεχνοτροπία ε, τέχνης, ξέρετε είναι κάποιοι τείχοι ας πούμε στις οποίες ε, ζωγραφίζουμε παράθυρα και νομίζουμε ότι είναι πραγματικά. Πολλές φορές ε, υπάρχει κάτι τέτοιο στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες των εθνικών κοινοβουλίων δείχνουν ότι κάτι κάνουν. Ενώ δεν το κάνουν οι βουλευτές, το κάνουν οι υπάλληλοι. Ε, δείχνουν ότι το σύστημα αυτό ε, είναι περίπλοκο της ε, πρόορης προειδοποίησης, έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά κάτι καταφέρνουν και σε σχέση με αυτό. Και αυτό ισχύει και για το διάλογο ανάμεσα στα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, που είναι ένας διάλογος κοφών μερικές φορές. Παράδειγμα, οι σημερινές διαπραγματεύσεις, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το διακοινοβουλευτικό φόρουμ του άρθρου 13. Την προηγούμενη εβδομάδα οι κανόνες λειτουργίας για το φόρουμ αυτό έγιναν αποδεκτοί με πάρα πολύ κόπο και δεν είμαι βέβαιος μετά από δύο χρόνια διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, δεν ομιλώ εδώ σαν ε, επιστήμονας αλλά σαν πολίτης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ αρνητικό που χρειάστηκαν δύο χρόνια για τους διαδικαστικούς κανόνες. Νομίζω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση οι πολιτικοί δεν βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων και θα πρέπει να είναι δυνατόν στο Εθνικό Κοινοβούλιο να ελαφρύνει λίγο τον τρόπο με τον οποίο ελέγχει και τα δημοσιονομικά. Thank you very much, ε, Professor. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Ρόζενμπεργκ. Τελευταίος ομιλητής ε, σήμερα ο κ. Φιλίππο Αχιέ από τη Βουλή του Λουξεμβούργου είναι ε, επικεφαλής του Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και για την πρόσκληση. Μπορούσαμε να περάσουμε στις πρώτες διαφάνειες. Ε, θα χωρίσω σε τέσσερις ενότητες το θέμα μου. Να θυμίσω μια επισκόπηση σύντομα ε, τις εργασίες που έχουν γίνει. Δεύτερον, συνθήκες, τα εθνικά κοινοβούλια. Τρίτον, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε την οικονομική διακυβέρνηση και τα εθνικά κοινοβούλια. Και μια τέταρτη ενότητα, να δούμε πώς έχουν οι διάφορες προτάσεις σήμερα για τη βελτίωση ε, της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Γενικά, όταν γίνεται λόγος για αυτονομία, για κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι πολλά στοιχεία θα πρέπει να έχουμε διάφορα πράγματα στο μυαλό μας και μεταξύ αυτών πώς ορίζεται η νομοθετική ατζέντα, η νομοθετική δουλειά αυτή καθ' αυτή και η κοινοβουλευτική και βεβαίως ο έλεγχος για τον προπολογισμό και ε, γενικότερος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Γενικά ε, στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για αποκοινοβουλευτικοποίηση του ρόλου των κοινοβουλίων στις 28 δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ε, η νομοθετική και η πολιτική ατζέντα για διάφορους λόγους ε, είναι στα χέρια κυρίως των κυβερνήσεων. Και στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ένα στοιχείο ενδεικτικό για το γεγονός ότι εκφεύγει η πολιτική ζωή του κοινοβουλευτικού ελέγχου και είναι στα χέρια των κυβερνήσεων. Πού οφείλεται αυτό. Υπάρχουν νέες μορφές συντεχνιών ε, είναι νέα μορφή διακυβέρνηση οικονομικής και νομισματική. Οι ε, κυβερνήσεις έχουν διάφορες επιτροπές εμπειρογνωμόνων, συμβουλευτικές που τι πλαισιώνουν και όλο και περισσότερο γίνεται εξωτερική αξιολόγηση των κυβερνητικών πολιτικών, ακόμα και της δημοσιονομική πολιτική του προπολογισμού δηλαδή. Έχουμε κατακαιρματισμό των διαφόρων φορέων και το Κοινοβούλιο είναι πλέον ένας φορέας μεταξύ πολλών άλλων. οι ε, κυβερνήσεις έχουν τους τεχνοκράτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε ιδιωτικοποίηση της αξιολόγησης των δαπανών και ε, γενικά διάφορες δομές που ξεφεύγουν από το Κοινοβούλιο. Τέσσερις είναι οι βασικές ε, αποστολές του Κοινοβουλίου να ε, κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο, να κάνει διάλογο με τα θεσμικά όργανα, να ελέγχει με βάση την επικουρικότητα αυτό που αναφέραμε προηγουμένως και να ε, προχωρεί σε κοινοβουλευτική συνεργασία με άλλα κοινοβούλια. Αν δούμε λοιπόν το σύνολο των συνθήκων από τη συνθήκη του Μαστρίχτ και μετά, τα εθνικά κοινοβούλια, κατ' εικόνα θα έλεγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν ε, μια διαδικασία πολύ βαριά, πολύ βραδία, ατέρμονη, με κολυσίεργιες στη λήψη των αποφάσεων. Και αυτό που μπορεί στη συνθήκη της Λισαβόνας να φάνηκε ως πρόοδος, ε, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, διαφωνώ με τους συναδέλφους. Οι διάφορες ε, συνθήκες και τα σύμφωνα μάλλον για την οικονομική διακυβέρνηση έχουν μειώσει το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων σε σχέση με εκείνο που είχαν πετύχει από τη ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως θύμισε και ο φίλος Ρόζεμπεργκ, υπάρχει διαφορετικός έλεγχος από κοινοβούλιο σε κοινοβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη ετερογένεια στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο οι εθνικές βουλές. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει διακοινοβουλευτική συνεργασία, γιατί τα εθνικά κοινοβούλια δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουν τι ίδιε εξουσίε, δεν έχουν τι ίδιες παραδόσεις, δεν έχουν την ίδια ιστορία, δεν έχουν το ίδιο όραμα για τα ευρωπαϊκά δρόμενα. στην πανεπιστημιακή συζήτηση προβληματίζει τους ειδικού ε, η συνδίκη της Λισαβόνας. Ε, αυτή στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταρρύθμιση και θεσμική και δημοκρατική ήταν μια αφετηρία ή ένα τέρμα. Έχει ολοκληρωθεί μια προσπάθεια ή αρχίζει τώρα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τα γνωρίζετε όλα αυτά, αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 12 ορίζει ε, διάφορες ε, ε, αρμοδιότητες και αναγνωρίζει εξουσίες για τα εθνικά κοινοβούλια. Και στη συζήτηση που γίνεται υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το ε, ποια είναι η πραγματική εμβέλεια της συνθήκη της Αβώνα. Ορισμένοι θεωρούν ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν περισσότερο ρόλο στην εθνική επικράτεια από ότι στην ευρωπαϊκή. Αυτό θα ήταν ένα παράδοξο, γιατί μια Ευρωπαϊκή Συνθήκη επιτρέπει στα Εθνικά Κοινοβούλια να ελέγχουν περισσότερο τις κυβερνήσεις του από ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης, δεν συζητείται καθόλου τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται οι ευρωπαϊκές ε, οδηγίες σε εθνικό επίπεδο, που είναι κατά κύριο λόγο η ευρωπαϊκή δουλειά που κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίση, τι γίνεται με τον έλεγχο τη επικούρικότητα και με ποιο τρόπο ασκείται αυτό από το κοινοβούλια. Όλοι αυτοί είναι προβληματισμοί και ερωτηματικά. Βεβαίω μπορεί να υπάρχει αναγνώριση των ε, διαφόρων μορφών συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων, κατοχυρωμένη αυτή στη συνθήκη της Λισαβόνα, αλλά συνήθως γίνεται αυτή με τρόπο άτυπο. Ακούσαμε προηγουμένως ότι χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια για να δούμε με ποιο τρόπο θα λειτουργεί το διακοινοβουλευτικό φόρουμ. Αυτή όμως η άτυπη συνεργασία είναι εις βάρος ε, της ε, δραστηριότητας και των εργασιών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει λοιπόν να επισημοηθεί πολύ περισσότερο και να κατοχυρηθεί στις επόμενες μεταρρυθμίσεις και να θεωρήσει των συνθήκων μια επίσημη τυπική συνεργασία και όχι άτυπη μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων. Προχωρούμε κάποιες ε, διαφάνειες πιο κάτω. Για τον έλεγχο της επικουρικότητας τελικά τι διαπιστώνουμε. Ότι μόλις 10 με 15% από το 2010 του συνόλου των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησαν σε έλεγχο της επικουρικότητας. Αυτό μπορεί να είναι κάτι καινούριο και δύσκολο να θεσπιστεί, αλλά είναι πολύ ισχνός αποτέλεσμα. 10 με 15%. Επόμενη διαφάνεια. Το 2014 είχαμε μια μικρή υποχώρηση και θα το αναγνώριζε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ήταν προς το τέλος της θητείας της η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν έκανε πολλές νομοθετικές προτάσεις και δεν χρειαζόταν και μεγάλο έλεγχο από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όπως είπε ε, ο συνάδελφος προηγουμένως, τα κοινοβούλια από τις σκανδιναβικές χώρες έχουν υπερεκπροσώπηση στον έλεγχο της επικουρικότητας. Αυτό οφείλεται σε μια συστηματική ε, άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για όλες τις οδηγίες. Αυτό όμως που επίσης διαπιστώνουμε είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες όταν κάνουν αυτό τον έλεγχο της επικουρικότητας και χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Οι ετελογημένες νόμες καμιά φορά ερμηνεύουν την αρχή της επικουρικότητας με πολύ ευρύτερο τρόπο από ότι το ίδιο το πρωτόκολλο της συνθήκης. Και επίσης υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων για την εφαρμογή και την εκτέλεση της αρχής της επικουρικότητας. Άρα δεν έχουν όλοι τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, ούτε προσθέτουν την ίδια σημασία στον έλεγχο επικουρικότητας και στα αντίστοιχα κριτήρια. παραμένουμε σε επίπεδο πανεπιστημιακών ακαδημαϊκών συζητήσεων για την επικουρικότητα, ο νέος μηχανισμός μπορεί να έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου, αλλά δεν είναι βέτο. Ούτε είναι επιθυμητό κάτι τέτοιο, ε, ούτε δυνατότητα αναστολής μιας απόφασης. Τώρα, όχι οι πολιτιολόγοι, αλλά οι νομικοί θεωρούν ότι ο έλεγχο τη υποκριτικότητα είναι μια επινόηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και είναι κάτι το οποίο χρησιμεύει περισσότερο στι κυβερνήσει από ό,τι στα κοινοβούλια τα ίδια. Συνέχεια, πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να μπω σε όλε τι λεπτομέρειε. Μπορείτε να διαβάσετε τις διαφάνειες στη συνέχεια. Αν δούμε λοιπόν τις διάφορες συνθήκες και τα σύμφωνα που εγκρίθηκαν από το 2009 για την δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση, βλέπουμε μια πρώτη δυσκολία. Αυτά τα σύμφωνα και οι συνθήκες εντάσσονται ταυτόχρονα και στη διακυβερνητική μέθοδο και στην κοινοτική. Ορισμένα μάλιστα είναι πιο κοντά στην διακυβερνητική μέθοδο. Αυτό έρχεται να δυσκολέψει τη δουλειά των Εθνικών Κοινοβουλίων στην οικονομική και δημοσιονομική τους διακυβέρνηση. Ας αφήσουμε στην άκρη όλες τις συνθήκες και την ανάλυση τους θέλω να πω κάτι γενικά για τη διακυβέρνηση και όλα τα σύμφωνα της οικονομικής διακυβέρνησης και της δημοσιονομικής. Πρώτον, σταδιακά, και λυπάμαι που το λέω, βλέπουμε να αποσυνδέεται ο προπολογισμό από τα κοινοβούλια για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι στη τελευταία συνθήκη και το τελευταίο σύμφωνο για την σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση, που είναι διακυβερνητική, το βασικό στοιχείο και ο άξονας του συμφώνου είναι η σύνοδο κορυφή της Ευρωζώνης, δηλαδή η αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων των μελών ε, της Ευρωζώνης. Το οποίο όμως, όργανο αυτό, ε, ουσιαστικά ε, διαφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου των εθνικών κοινοβουλίων. Ενισχύει το ε, ορθολογικό κοινοβουλευτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως. Και οι διάφοροι μηχανισμοί που έχουν ε, δημιουργηθεί μειώνουν ή περιορίζουν τον παραδοσιακό ρόλο των κοινοβουλίων στον έλεγχο της εκτέλεσης του προπολογισμού. Εντάξει, είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι έχουν συσταθεί διάφορα συμβούλια για τις κυβερνήσεις ε, στα πλαίσια των συμφώνων σταθερότητας και ανάπτυξης Τα συμβούλια αυτά σπανίως έχουν σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Προχωρώ αρκετές διαφάνειες πιο κάτω και έρχομαι τώρα στο πλαίσιο των προτάσεων στην περιγραφή της κατάστασης και στα συμπεράσματα. Αν δούμε λοιπόν τις διάφορες προτάσεις για τη βελτίωση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, παρατηρείται πολύ μεγάλη δραστηριότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων για να βρεθούν νέοι τρόποι ε, για να συνδεθούν καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Έκθεση ε, του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, έκθεση ε, του Κοινοβουλίου της Δανίας, Κόζακ και η μελέτη της Βρετανικής Βουλής των Λόρδων συγκλίνουν ε, όλες αυτές οι εκθέσεις ως προς το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και έναν ανταγωνισμό μεταξύ των κυβερνήσεων. Στην έκθεση, ας πούμε, της ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, που πρόσφατα δημοσιεύτηκε. Είναι πολύ μεγάλες οι αποκλήσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και της δράσης και των δραστηριοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων για να αναβαθμίσουν το ε, ρόλο τους. Μερικά Δύο-τρία παραδείγματα μόνο και μετά θα καταλήξω. Όλη η συζήτηση αυτή που γίνεται για την πράσινη κάρτα ε, και ξεκίνησε στην Κόζακ δείχνει πόσο αμφίσιμη είναι η κατάσταση. Από τη μια, ορισμένα κοινοβούλια μέχρι που αδιαφορούν για την ε, πράσινη κάρτα αυτή. Αλλά θέλουν, επιθυμούν διακαώς ε, την πράσινη κάρτα αυτή. Αν δούμε όμως τις διαφορετικές θέσεις, όταν γίνεται λόγος για την πράσινη κάρτα δεν εννοούν όλα τα κοινοβούλια το ίδιο πράγμα και ταυτόχρονα κάνουν, μάλλον έχουν πολύ μεγάλη συνένεση ε, ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει πάρα πολλές εξουσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα κοινοβούλια. δυσκολία είναι ότι κατακλείζονται από πληροφορίες και τελικά δεν μπορούν να κάνουν την κοινοβουλευτική τους δουλειά σωστά. Ε, συμφωνούν σε αυτό όλες οι εκθέσεις. Ένα ακόμα στοιχείο, πολύ ενδιαφέρουσε όλες αυτές οι μελέτες και εκθέσεις, υπάρχει απόλυτη και μόνιμη επιθυμία για συστηματική συνεργασία μεταξύ ε, των μελών της, και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και λογοδοσία των κυβερνήσεων ε, απέναντι στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Φτάνω, προχωρώ προς τα συμπεράσματα. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που απορρέει από όλε αυτές τις εκθέσει είναι ο ρόλος των ίδιων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει και εδώ ευρεία συναντήληψη για το εξή γεγονό. Θα πρέπει να υπάρχουν λιγότερε ειδικέ ευρωπαϊκές επιτροπές ε, και περισσότερη ευρωπαϊκή διάσταση στι επιμέρου επιτροπέ, μεταφορών, ε, εμπορίου ε, ε, κτλ. Γεωργίας ή όποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Να μην ασχολούνται δηλαδή με τα ευρωπαϊκά θέματα μόνο οι επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων. Και έρχομαι στο τελευταίο θέμα, στην τελευταία διαφάνεια. Είναι πολύ μεγάλη, λοιπόν, είπαμε η ετερογένεια των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε μείωση του ρόλου των κοινοβουλίων και δυσκολεύεται η ε, επίτευξη κοινών ε, στόχων και στρατηγικής για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Επίσης, οι συνθήκες και ιδιαίτερα οι συνθήκη της Λισαβόνας έχουν μία ε, νομική τύπο λατρεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα δικαιώματα που δίνουν. Δίνουν νέα δικαιώματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα ασκήσει κανείς. Ιδιαίτερα λοιπόν τα σύμφωνα ε, για τα οικονομικά ε, έχουν ε, απελευθερώσει τις κυβερνήσεις από τις ευθύνες τους απέναντι στα εθνικά κοινοβούλια και δημιουργείται ένα δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο δεν έρχεται να καλύψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Και επίσης πρέπει να γίνει πολύ σημαντική δουλειά για να δούμε πώς μπορούν να ενισχυθούν τα εργαλεία και τα μέσα για τα, όλα τα κοινοβούλια στον έλεγχο της οικονομικής διακυβέρνησης. Πολύ δε περισσότερο που υπάρχει ε, διαίρεση μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται τέτοιος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ενώ οι κυβερνήσεις έχουν ε, ε, ξεκάθαρα στο μυαλό τους ποιες είναι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και προηγούνται πολύ στην προσπάθεια αυτή, ενώ τα κοινοβούλια υπολείπονται κατά πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, ε, έχουμε τώρα αυτές τις γαλάζιες κάρτες και θα ήθελα να εξηγήσω και στους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων ότι στις ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται συζήτηση. Δηλαδή δεν καλούμε μόνο εμπειρογνώμονες για να τους ακούσουμε, αλλά γίνεται και συζήτηση ε, και διάλογος και βεβαίως στο τέλος της ακρόασης απαντούν ή αντιδρούν οι εμπειρογνώμονες. Παρακαλώ λοιπόν να λάβετε το λόγο και να κάνετε μόνο τοποθετήσεις. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες, γι' αυτό τους καλέσαμε. Ο Τούρκος συνάδελφος, ο κύριος Κιουτσούκ Τσάν, έχει πρώτο το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρέμβασή μου θα είναι σύντομη και θα κάνω μια ερώτηση. Ε, στις παρουσιάσεις εστιάσαμε στα, στο θεσμικό επίπεδο και στα μέσα που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω όμως πως λείπει ένα στοιχείο, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογέ. Στις τελευταίες ευρωεκλογέ, αν θυμάμαι καλά, η συμμετοχή ήταν περίπου 42,5%. Αλλά και στις εθνικές εκλογές, αν κοιτάξουμε την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούμε μια παρόμοια τάση. Μειώνεται το ενδιαφέρον για την πολιτική, μειώνεται η συμμετοχή στα κοινά και αυτό αναρωτιέμαι αν είναι ένας, ε, μια ένδειξη για την έλλειψη εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα από τους πολίτες της Ένωσης σε πολλές χώρες. Και πιστεύω πως αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν κάνουμε λόγο για λογοδοσία, για διαφάνεια και για τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορούν οι πολίτες να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη. Μπορεί η Ευρώπη να γίνει πιο ορατή, γιατί αυτό που λείπει είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτή τη στιγμή ε, πάσχει και πρέπει να απασχολήσει αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η ερώτησή μου σχετίζεται άμεσα με αυτό. Αναρωτιέμαι αν οι εμπειρογνώμονες έχουν εξετάσει αυτήν την πτυχή και την έχουν αναγνωρίσει ως κάτι που λείπει από την ε, ανταλλαγή απόψεων. Αυτή δηλαδή η άμεση δημοκρατία, αυτή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Μπέρτσαου από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω πως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αποφασιστική σημασία μάλιστα, να ενισχυθεί ο διακοινοβουλευτικό διάλογο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Στην ε, Ρουμανία έχουμε ειδική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Κοινοβούλιο και εκεί δεν συντάσσονται μόνο γνωμοδοτήσει οι οποίες ε, αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και κάθε μήνα έχουμε ώρα των ερωτήσεων για ευρωπαϊκά ζητήματα. Για παράδειγμα, για τη μετανάστευση, το σχέδιο Juncker, τη μεταναστευτική πολιτική, το ψηφιακό θεματολόγιο, την Ενεργειακή Ένωση και μου έκανε μεγάλη έκπληξη λοιπόν ε, αυτό που άκουσα από τον ε, κύριο Ρόζενμπεργκ, ο οποίος είπε ότι το κοινοβούλιο στη Ρουμανία δεν ανήκει στα ενεργά και τα δραστήρια κοινοβούλια. Η τελευταία ε, ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι η Βουλή της Ρουμανίας βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Γι' αυτό ίσως ε, καλό θα ήταν να συμβουλευτούμε πιο πρόσφατα στοιχεία. Στη Ρουμανία λοιπόν Υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθεσία σχετικά με την συνεργασία Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης. Η συνεργασία στην αρχή είχε κάποια προβλήματα, όμως τώρα όλα πάνε μια χαρά και ο κοινοβουλευτικός ε, έλεγχος στα ευρωπαϊκά ζητήματα ασκείται επαρκώς. Η Προεδρία λοιπόν είναι επίσης δεσμευμένη να ενημερώνει συνεχώς. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι παράγραφοι 9 και 10 με ανησύχησαν κάπως και θα ήθελα να σας ατονίσω την προσοχή, την, να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι τα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν εξετάζονται μόνο από την κυβέρνηση, πρέπει να εξετάζονται γενικότερα από το Κοινοβούλιο. Έπειτα, αυτό ισχύει και για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών ε, δομών. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έπρεπε να ελέγχουμε, για παράδειγμα, τις ε, διαπραγματεύσεις ε, για την Ευρωπόλη, το τι γίνεται, τις εξελίξεις. Και επίσης χρειάζεται στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε η συνεισφορά των εθνικών κοινοβουλίων να λαμβάνεται υπόψη. Ε, από ε, πλευράς επικουρικότητας τώρα, να σας πω ότι πιστεύω πως θα ήταν ίσως καλό να έχουμε ένα σύστημα βέλτιστων πρακτικών, δεν νομίζετε. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Διότι χρειάζεται επίσης και επαρκής ε, χρόνος για να μπορέσουμε να εξετάσουμε σε κάθε την κάθε πρόταση που μας θέλει η Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή το περιθώριο είναι 8 εβδομάδες και δεν μας φτάνει. Και έπειτα, πιστεύω πως χρειάζεται και ένας έλεγχος της συνέχειας, μια παρακολούθηση της κάθε δράσης. Πιστεύω πάντως πως εδώ αυτή τη στιγμή κάναμε μια συζήτηση σε βάθος, αλλά θα ήθελα να ελπίζω ότι θα συνεχίσει αυτό και θα γίνει πράξη. Η συνεισφορά λοιπόν των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πιστεύω πολύ σημαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Το βασικό μήνυμα από τις συζητήσει σήμερα το απόγευμα και το πρωί είναι ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ουσία και όχι επικορικότητα. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι η ευκαιρία των κοινοβουλίων να κοιτάξουν το περιεχόμενο των προτάσεων και όχι να ξοδεύουν όλοι τους την ενέργεια σε θέματα ελέγχου της επικουρικότητας. Στην ουσία η επικουρικότητα σπάνια αποτελεί πρόβλημα. Μπορεί να χρειάζεται να λειτουργήσει σαν αγγίηση, αλλά από την άλλη μετά από έξι χρόνια που έχει δημιουργηθεί ο, ο μηχανισμός αυτός έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο δύο φορές ε, ε, και για την πορτοκαλί κάρτα δεν έχει υπάρξει τέτοια αντίστοιχη περίπτωση. Γι' αυτό και προσέχει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγουν ορισμένοι τις προτάσεις της λόγω της ύπαρξης της επικουρικότητας, γιατί όχι. Αλλά κυρίως γιατί όσο περνάει ο χρόνος, ένας ένα αυξανόμενος αριθμός νομοθετικών προτάσεων της Ένωσης οδηγούν στην τροπολόγηση της υπάρχουσας τροπολογίας και όχι σε νομοθεσία σε νέους τομείς. Αυτό είναι φυσιολογικό, να αλλάζουν δηλαδή τα στοιχεία αυτά. Και όταν μιλάμε για την αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε αν πράγματι η εθνική αυτή νομοθεσία ή η υπάρχουσα γενικά νομοθεσία επαρκεί. Σε όλα τα επίπεδα κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την ε, ειδική πλειοψηφία, το 65% δηλαδή εφόσον χρησιμοποιήσουμε και την πληθυσμιακή στάθμιση, των υπουργών που είναι υπόλογοι ε, στα δικά τους κοινοβούλια αλλά αποφασίζουν στο Συμβούλιο. Το τίμημα λοιπόν της παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας μειώνεται γιατί απαιτείται η πλειοψηφία των κυβερνήσεων που θα πρέπει να στηρίξει την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι δεν χρησιμοποιείται η βασική αυτή αρχή. Πώς μπορούν λοιπόν τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια να επηρεάσουν την ουσία της νομοθεσίας και όχι να ανησυχούν για θέματα επικουρικότητας. Μέσω διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω επίσης συζήτησης με τον αρμόδιο υπουργό πριν πάει στις Βρυξέλλες, προκαταρπτική δηλαδή επεξεργασία. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο θα κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια, δεν θα τους πει το ευρωπαϊκό επίπεδο που θα τους κάνουν. Αλλά μέσα σε όλα αυτά και λέγοντας ότι συνήθως η επικουρικότητα δεν είναι πρόβλημα, Τώρα έχουμε έναν πρωθυπουργό που ζητάει κόκκινη κάρτα. Εγώ λέω ναι, να έχουμε κόκκινη κάρτα, δεν είναι πρόβλημα γιατί δεν θα υπάρξουν προτάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κόκκινη κάρτα, θα ήταν πάρα πολύ σπάνιο. Θα μπορούσαμε να το δεχθούμε αυτό, έτσι ώστε αν είναι απαραίτητο τότε να μπλοκάρει κανείς μια διαδικασία αν παραβιάζει την επικορικότητα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποσύρει την πρότασή της όταν φτάνει στο επίπεδο ας πούμε της πορτοκαλί κράτας. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα, Κόρμπετ. Νομίζω ότι η βασική ιδέα είναι η διεύρυνση, ε, θα έλεγα, της ιδέας, της αρχής της επικουρικότητας. Υπάρχουν πολλά θέματα στο μέλλον που μπορεί να καλυφθούν από την πρόταση αυτή, όπως η αιρεσιμότητα. Θα δούμε, αυτό είναι θέμα συζήτησης, λέει ο Κόρμπετ. Στα Ολλανδικά θα μιλήσω και πάλι. Πρώτον, θα ήθελα να πω στον συνάδελφο από την Τουρκία ότι ήμουν επιμακρών εισηγήτρια για την Τουρκία. Και όταν πρέχεις από μία χώρα που υπάρχει τέτοια πόλωση, τότε είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου είναι κάπως πιο ήπιες οι δημοκρατίες και πιο έξυπνες. Επίσης θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα κατόφλια για να μπει στη Βουλή. Στην Τουρκία είναι γύρω στο 10%. Μήπως έχει και αυτό σχέση και είναι πιο πολιτικοποιημένος ο κόσμος και ψηφίζει. Δεν ξέρω, λέω. Ε, πρόεδρε, το σημερινό θέμα ποιο είναι τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ε, για την επικουρικότητα. Προσωπικά πιστεύω ειλικρινά ότι το πρόβλημα δεν είναι η επικουρικότητα και συμφωνώ με τον Ρίτσαρτ Κόρμπετ και θέλω να απευθυνθώ και στον, ε, ε, στον ειδικό μας από το Λουξεμβούργο που μας τα περιέγραψε πολύ μελανά τα πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ θυμάμαι τη συνθήκη του Μαστρίχ στη δεκαετία του 90 που είχαμε εδώ ένα κοινοβούλιο χωρίς αρμοδιότητες. Ήμουν βουλευτής τότε. Ένα τμήμα των αρμοδιοτήτων ε, προσθέθηκε αργότερα. Θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, Πρόεδρε, η επικουρικότητα ε, και ε, η έλεγχη που έχουμε για αυτήν πρέπει να μεταξελιχθεί Υπάρχει ένα πρόβλημα στα κράτη-μέλη. Δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο πολλές φορές της ε, νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Δεν συμφωνούν διότι ε, βρίσκουν ότι είναι υπερβολικά αναλογική για τη χώρα τους. Ε, θα πρέπει εκεί να γίνουν οι συμφωνίες και οι συζητήσεις. Και θέλω να πω κάτι στη συνάδελφο από την Ολλανδία και στον κύριο από τη Γαλλία. Έχετε εξετάσει και ερευνήσει τι γίνεται με κοινοβούλια, εθνικά μιλάω, όπου συνεργάζονται πολύ περισσότερο οι ευρωβουλευτές με τους εθνικούς βουλευτές. Παράδειγμα, στην Ολλανδία οι ευρωβουλευτές καλούνται, προσκαλούνται συχνά στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, πηγαίνουν στη Χάγη, μιλούν πέντε λεπτά και την υπόλοιπη ώρα κάθονται και ακούνε. Ε, υπάρχουν χώρες που δεν ε, το χρησιμοποιούν αυτό, αλλά στη Γερμανία έχουν και κοινέ μικτές επιτροπές κοινοβουλευτικές και στη Γαλλία είναι πολύ πιο στενός ο διάλογος ευρωβουλευτών με τους βουλευτές της Γαλλικής Συνέλευσης. και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει για να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκα το πρωί, το μακρύ χέρι της καταπολέμησης της, δημοκρα... ε, της ε, γραφειοκρατίας. Συγγνώμη. Αυτές τις ερωτήσεις είχα να κάνω. Ευχαριστώ τελείως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ατσιώτη Διτσέλτα από την Ιταλία. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που έχει εφαρμόσει αν θέλετε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων. Η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάζεται πριν από κάθε Συμβούλιο και να αναφέρεται επίσης στην έκβαση του Συμβουλίου εκ των υστέρων. Ταυτόχρονα στη διαδικασία διαμόρφωσης της θέσης υπάρχει μια υποχρέωση εμπλοκής του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα οι θεσμικές αλλαγές οι οποίες είναι υποσυζήτηση δεν έχουμε φτάσει παρά στον τελευταίο γύρο βέβαια αύριο μάλλον θα ξεκινήσει ο τελευταίος γύρος για πρώτη φορά προβλέπεται και στο Σύνταγμα η εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην ανάλυση και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Προβλέπεται επίσης και η αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο ε, της τελικής απόφασης γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Η εμπειρία λοιπόν την οποία έχουμε στο Κοινοβούλιο είναι ότι οι συζητήσεις και ο τρόπος με τον οποίο το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει την κυβέρνηση πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως και οι συζητήσεις τις οποίες έχουμε εκ των υστέρων, φαίνεται πολύ συχνά να φορούν γενικότερα θέματα σχέσεων της Ιταλίας ή της κάθε χώρας με την Ευρώπη σε επίπεδο συνολικότερο πολιτικών και υπάρχει θα έλεγα μία έλλειψη ανάλυση σε βάθος. Η κυβέρνηση τίνει να παρουσιάζεται με συγκεκριμένα περιορισμένα στοιχεία ενημέρωσης και η συζήτηση που ακολουθεί πάρα πολύ σπάνια ασχολείται με τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου θέματος. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν η πρότασή μου ή μάλλον η ερώτησή μου είναι αν κάτι τέτοιο συμβαίνει και με άλλα κοινοβούλια ή μήπως υπάρχουν περιπτώσεις με τις αφορμές των μεγάλων συμβουλίων οι συζητήσεις που κάνετε στα κοινοβούλια σας είναι πιο λεπτομερείς από τη δική μας. Λοιπόν, υπάρχει μια εμπλοκή επί της ουσίας σε επίπεδο γενικών στρατηγικών. Πάρα πολύ σπάνια υπάρχει λεπτομερής προετοιμασία. Και δεν ξέρω λοιπόν αν τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται ως κατεπήγοντα κάθε φορά και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν δυνατότητες εμπλοκής βαθύτερης. Δεν ξέρω αν σε ακαδημαϊκό επίπεδο μπορεί να υπάρξουν προτάσεις. Ο κύριος Χαουρέγγι από την Ισπανία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιρρογνώμονές μας για τις εκθέσεις για τις παρουσιάσεις τους. Νομίζω ότι ανέπτυξαν όλο το φάσμα των θεμάτων, την επικουρικότητα, τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου. Έχω τρεις ερωτήσεις να τους κάνω. Πρώτον, όταν εξετάσατε τις ε, κοινοβουλευτικές συζητήσεις στις παραμονές των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Δεδομένου ότι τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Σύνοδοι Κορυφή τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τεράστια σημασία μέχρι που κυριάρχησε η διακυβερνητική διάσταση επί της κοινοτικής θεώρησης της Ένωσης. Έχω λοιπόν την εξή ερώτηση. Γιατί με έχει προβληματίσει το γεγονός ότι ορισμένα κοινοβούλια δίνουν συγκεκριμένη γραμμή στις κυβερνήσεις, στις παραμονές των συμβουλίων. Αυτή η εντολή, η απόλυτη, δεν συνάδει με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία πάντα. Υπάρχουν πολλά τέτοια κοινοβούλια που δίνουν συγκεκριμένες εντολές στις κυβερνήσεις τους εν ώψη το Συμβουλίο, γιατί αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ε, προβληματικό και οδηγεί ε, σε ε, διατάραξη της λειτουργίας του Συμβουλίου. Κάνατε πολύ ωραίες ε, στατιστικές και μετρήσεις για όλες τις συνεδριάσεις που γίνονται κτλ. Τι γίνεται τώρα με τις συζήτηση μετά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Στα Εθνικά Κοινοβούλια λοιπόν. Μήπως εθνικοποιούνται εντός εισαγωγικών οι συζητήσεις. Δηλαδή αντί να συζητούν για την Ευρώπη σχεδόν όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια μεταφέρουν την ευρωπαϊκή συζήτηση και την ανάγουν σε εθνικά θέματα και αφήνουν την ευρωπαϊκή συζήτηση εκτός για διάφορους λόγους πιέσεων τοπικών, εθνικών, επικαιρότητα κλπ. Ε, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Και μια τρίτη ερώτηση. Ποιος ο ρόλος των περιφερειακών κοινοβουλίων σε χώρες αποκεντρωμένες. Παράδειγμα, η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει πολύ καλή πρακτική ε, στον τρόπο με τον οποίο εξετάζει την επικουρικότητα. Πώς συμμετέχουν λοιπόν οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατηδίων της Γερμανίας και τα κοινοβούλια των ομόσπονδων κρατηδίων. Γιατί αυτές οι τοπικές κυβερνήσεις στη συνέχεια καλούνται να εφαρμόσουν ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο Μάρκ Άνζελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με μια ερώτηση προ ε, την κυρία Νόιχολτ. Μα αναφέρατε τι διαφορετικέ διαδικασίε που ακολουθούν τα εθνικά κοινοβούλια ε, για να ελέγξουν την εκτελεστική του εξουσία. Φυσικά και χαρακτηρίζεται αυτό και από την ε, πολιτισμική διαφορά που υπάρχει από χώρα σε χώρα. Αλλά τι, τι είναι περισσότερο, οι πολιτισμικές διαφορέ, οι θεσμικέ διαφορέ, τι δημιουργεί αυτέ τι διαφορέ. και δεν θα έπρεπε ίσω να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στα εθνικά κοινοβούλια μεταξύ τους για να βελτιώνονται. Έπειτα, Αναφέρατε επίσης ε, και την εκ των προτέρων πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην κυβέρνηση. Μετά την ε, Προεδρία μας ε, θα κάνουμε μια αξιολόγηση της κατάστασης, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να είμαστε καλά ε, προετοιμασμένοι. Το προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά την μια συνεδρίαση του Συμβουλίου. Πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το διοικητικό προσωπικό λοιπόν, όπως αναφέρατε και εσείς κυρία Νόιχολτ. Ε. Καθηγητά Ρόζεμπερκ, ε, είπατε περίπου σχετικά πράγματα με αυτά που είπα εγώ σήμερα το πρωί, το mainstreaming, δηλαδή ένταξη των ευρωπαϊκών θεμάτων ε, στι ε, ε, γενικέ πολιτικέ. Έρχομαι στι Βρυξέλλε και διαπιστώνω ότι είμαστε μια μικρή ελίτ στην κάθε Εθνική Βουλή που ασχολούμαστε με ευρωπαϊκά θέματα. Γι' αυτό στο Λουξεμβούργο θελήσαμε να μην έχουμε μία Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ενταγμένοι και μοιράζονται τα διάφορα θέματα στη συνέχεια στις επιμέρους επιτροπές για να υπάρχει ακριβώς μια τέτοια εγκάρσια συζήτηση. Και χαίρομαι που αναφερθήκατε στη βράσινη κάρτα και είπατε ότι μπορεί να γίνει χωρίς τροποποίηση των συνθήκων. Και δεν πέσατε στην παγίδα όπως ορισμένοι που διαφωνούν με την πράσινη κάρτα που πιστεύουν ότι θέλουν να έχουμε εμείς ε, δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας ως Εθνικά Κοινοβούλια. Και μια ερώτηση προς τον καθηγητή ε, κύριο Πουαριέ. Ε, μιλήσατε για αποκοινοβουλευτικοποίηση. Μήπως είναι αυτό έλλειψη χειραφέτησης των κοινοβουλίων ή έλλειψη στράτευσης. Δεν είναι παρέτηση των κοινοβουλίων. Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Πώς το βλέπετε. Όταν μιλάω για χειραφέτηση, ε, θέλω να σας εξηγήσω το εξή. Δεν έγινε σήμερα, αλλά πολλέ φορέ έρχομαι στις Βρυξέλλες σε αυτές τις διακοινοβουλευτικέ συνεδριάσεις και βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοι από διάφορες χώρες, δεν θα τις κατονομάσω, που διαβάζουν ε, ομιλίες ε, τις οποίες έχω την αίσθηση έχουν γράψει τα Υπουργεία Εξωτερικών και όχι τα κοινοβούλια. Γι' αυτό μιλώ για χειραφέτηση των κοινοβουλίων από τις κυβερνήσεις. Αυτό θα βοηθήσει για να υπάρξει και καλύτερη συνεργασία μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και λοιπόν φορέων εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Mr. Duarte Κύριε Δουάρτε Duarte nesta intervenção gostava Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ μέρου τη ε, Βουλή τη Πορτογαλία ε, να εκφράσω τη στήριξή μα στην ε, πράσινη κάρτα. Πιστεύω πως χρειάζεται να φέρουμε το θέμα αυτό στην συζήτηση, αλλά και η πολιτική συζήτηση πρέπει να είναι και σχετική με τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Φυσικά η συζήτηση για ευρωπαϊκά θέματα έχει πολλές φορές λειτουργήσει εις βάρος της συζήτησης για τα εθνικά. Η Πορτογαλία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός καλού μαθητή. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων εξετάζει τις διάφορες προτάσεις, δεν έχει όμως την ευκαιρία και το χρόνο να διοργανώσει ανταλλαγή απόψεων ε, για θέματα που αφορούν τους πολίτες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν οι επιτροπέ αυτέ να μπορούν να συνεισφέρουν θετικά για του πολίτε. Όχι μόνο να υπάρχουν και να ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά να έχει και αποτέλεσμα αυτό. Επίση χρειάζεται να ενισχύσουμε την ε, αίσθηση των πολιτών μας ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Και επίσης πρέπει να φέρουμε κοντά τους λαούς της ε, Ευρώπης ε, πολιτισμικά. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει γενικότερα, όχι μόνο στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά πρέπει να αναζωοποιηθεί το ενδιαφέρον των ε, πολιτών για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χάνιγκαν από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ παρουσιάσεις και πραγματικά μου έδωσαν τροφή για σκέψη. Στηρίζω τις ε, προτάσεις για μεταρρύθμιση, στηρίζω και την πρόταση για την πράσινη κάρτα και τις ιδέες του Μαρκ Άγγελς. Πιστεύω όμως πως πρέπει να δημιουργηθούν ε, κριτήρια σχετικά με την επικουρικότητα. Τώρα, όσον αφορά τον έλεγχο, εμείς ε, υιοθετήσαμε το σύστημα του mainstreaming, της συνεκτίμησης δηλαδή στην ευρωπαϊκή πολιτική και ο έλεγχος αυτός μάλιστα συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι διαφορετικό δηλαδή σε σχέση με πριν. Αρχικούσαμε, επίσης για παρουσιάσεις ε, ευρωπαϊκών ζητημάτων στην Ολομέλεια των Εθνικών Κοινοβουλίων κτλ. Εγώ πρέπει να σας πω ότι κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο της ε, Ιρλανδίας έχει ε, μία τέτοια συνάντηση όπου εξετάζονται και στατιστικά στοιχεία και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν μία έντονη ενασχόληση του Εθνικού Κοινοβουλίου με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ακούμε τις ε, κριτικές, θετικέ και αρνητικέ και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ε, επιδόσεις μας ως ε, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων και ως Εθνικό Κοινοβούλιο γενικότερα. Με μεγάλο ενδιαφέρον επίσης άκουσα τις προτάσεις για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, υπάρχουν διάφορα προγράμματα ή ανά αναχώρα, ε, τα οποία ακολουθούμε και ε, δημοσιονομικά θέματα επίσης. Υπάρχουν και διάφορες προτάσεις για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω την άποψη των προσκεκλημένων σχετικά με τις προτάσεις αυτές και το κατά πόσο αυτές θα ενισχύσουν όντως τον ρόλο του Κοινοβουλίου τα δημοσιονομικά, στην κατάρτιση του προπολογισμού και να έχουν κάποιε δικέ του προτάσει για το τι χρειάζεται. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο Λόρδο Μπόσουελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχά ότι εγώ ίδιος ε, συνέταξα αυτά τα σχόλια, δεν τα έκανε άλλο για μένα. Προσπάθησα λοιπόν κάποια ε, από τα ε, όσα άκουσα να τα παρουσιάσω εδώ. Καταρχάς, το θέμα της προσοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως ε, πρέπει να προσέξουμε όταν διεξάγουμε ελέγχους να μην χάσουμε το στόχο. Πρέπει να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις, ε, τα αποτελέσματα της πολιτικής. Επίσης, ε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αναφορά στην πληθώρα των πληροφοριών. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε και πώς θα τη διαχειριστούμε και πώς θα ξεδιαλέξουμε την, ε, τα βασικά από τα λιγότερο βασικά. Έπειτα, είδα ότι υπάρχει μια τεράστια πολυμορφία εθνικών πρακτικών, όπως ε, έδειξαν οι διαφάνειες. Και αυτό φυσικά ε, συνεπάγεται και διαφοροποίηση πόρων από κοινοβούλιο σε κοινοβούλιο. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, πρέπει να είσαι ευέλικτο στην προσέγγιση σου. Επίσης υπάρχει και μεγάλη ε, πολυμορφία στα θέματα τα οποία απασχολούν το κάθε κοινοβούλιο. Ακούσαμε και για τις πράσινες κάρτες και αυτό είναι θέμα πρωτοβουλίας. Υπάρχει δηλαδή, ε, υπάρχουν οι δύο πλευρές του νομίσματος, η απορρίθμιση ή η συνέχεια, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και κάτι άλλο που ακούσαμε σήμερα το πρωί είναι ε, για τις ε, διαδικασίες ελέγχου και φυσικά αρμόδιοι να μιλήσουν γι' αυτό και να το κρίνουν είναι κυρίως το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύω. Ε, και τώρα, κύριε Κόρμπετ, είπατε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από αυτά. Ε, πρέπει σίγουρα να το εξετάσουμε αυτό και πρέπει να προβλέψουμε και κάποιε κυρώσει ενδεχομένω σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική. Είναι προφανέ επίση, ε, πιστεύω, το πώ διαχειριζόμαστε ε, την κατάσταση και είναι προφανές ότι, ότι χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια και εμείς εδώ μπορούμε να βάλουμε τα θεμέλια γι' αυτό χωρίς να διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία ή οι αρμοδιότητες των διάφορων και φυσικά α μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πολιτικό πλαίσιο, ότι το εκλογικό σώμα έχει και αυτό ε, ανάγκες ε, και αυτό επηρεάζεται από lobbying, από τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να είμαστε περισσότερο ευέλικτοι και ε, ταχύτεροι. Πρέπει να ακούμε τις ανάγκες των πολιτών και να τις εξυπηρετούμε. Χρειάζεται καταρχάς σε τεχνικό επίπεδο να δούμε πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα σε αυτές τις προτάσεις σε μία περιεκτική λύση. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο συνεργασίας θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα θέμα το οποίο θα εξετάσει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όταν ήμουν στην ε, Κάτω Βουλή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε ε, ένα θέμα που αφορούσε τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και σε αυτό συνεργάστηκαν ε, εκπρόσωποι από πολλά θεσμικά όργανα. Χρειάζεται επίσης να σκεφτούμε και πολιτικά, να σκεφτούμε για ε, την πιθανή δημιουργία ενός κοινοβουλευτικού χώρου που θα αποτελείται και από εθνικά κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες, θα έχει το δικαίωμα δηλαδή να συνεισφέρει ουσιαστικά στην νομοθετική διαδικασία. Και πρέπει να μην ξεχνάμε και την νομιμότητα. Πρέπει να συνηθίσουμε επίσης να συνεργαζόμαστε, διότι εάν καταφέρουμε να συνεργαζόμαστε θα οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια και κάποιες ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες. Μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων υπάρχει ένα του οποίου η ανεξαρτησία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και υπάρχει το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης του Ιδρύματος αυτού που δεν είναι υπεύθυνο μόνο για θέματα νομισματικής πολιτικής αλλά στα πλαίσια και της Τραπεζικής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη και για την εποπτεία των τραπεζών και θα ελέγξει ένα μεγάλο τμήμα του τρίτου πυλώνα, πιο πιθανό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναπτύσσουμε στην παρούσα φάση Εξετάζουμε τις ευθύνες λοιπόν της Κεντρικής Τράπεζας και προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να νομιμοποιήσουμε δημοκρατικά τις νέες αυτές δραστηριότητες. Καταλήξαμε σε διάφορες προτάσεις όπως η υπογραφή κάποιων μνημονίων κατανόησης, σε σχέση με τις δραστηριότητες της τράπεζας για τον έλεγχο διαδικασιών ας πούμε κλεισίματος τραπεζών ή ενίσχυσης διάσωσης τραπεζών. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής πρόκληση έβρεση της σωστή ισορροπίας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών υπέρ της ανεξαρτησίας των πιστοτικών ιδρυμάτων και του δημοκρατικού ελέγχου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια πάνω σε αυτό. Αν βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες εδώ ή μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο η δημοκρατική νομιμότητα μπορεί να γίνει αντικείμενο εγγύησης. Δεύτερον, πάρα πολύ συχνά οι συμφωνίες οι οποίες οδηγούν στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς σταθερότητας και επίσης στα διάφορα ταμεία είναι στην ουσία διεθνείς συμφωνίες οι οποίες ονομάζονται διακυβερνητικού τύπου συμφωνίες οι οποίες όμως παραμένουν θεωρητικά στα πλαίσια της συνθήκης και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαφοροποιείται σε σχέση με τη νομική τους βάση. Είναι λοιπόν θεμητό σε αυτή την περίπτωση καθαρής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας Είναι δικαιολογημένο λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές να περιμένει κανείς από τα κοινοβούλια και από το Εθνικό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ή μήπως θα έπρεπε να καταλάβουμε ότι τα δικαιώματα των κοινοβουλίων στην ουσία περιορίζονται όταν ξεπερνούν τις συνθήκες οι κυβερνήσεις και υπογράφουν διεθνείς συμφωνίες εκτός αυτών. Ξέρουμε γιατί το κάνουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Θα δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει από σας. Η κυρία Νόιχολντ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Είναι θετικό για μας τους πανεπιστημιακούς να βλέπουμε τον τρόπο που γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω έχει σχέση με τις δυνατότητες διαλόγου. Πολλές φορές η πολιτική δραστηριότητα και η έρευνα στα πανεπιστήμια δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη σχέση και αυτό δεν είναι καλό. Τώρα για την έλλειψη συμμετοχής στις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μας απασχολεί όλους. Και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Επιτροπή κτλ σχετικά με την προετοιμασία για τις εκλογές την προηγούμενη φορά ήταν κάτι το διαφορετικό. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η προσπάθεια έγινε αλλά παρόλα αυτά δεν απέδωσε. Βλέπουμε όμως πάρα πολλές διακυμάνσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ορισμένες χώρες ξέρετε ότι υπήρξαν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής. Μία από τις εξηγήσεις είναι που δίδουν και οι πανεπιστημιακοί και οι πολιτικοί επιστήμονες είναι η έλλειψη πολιτικής ε, συζήτησης, η έλλειψη πολιτικοποίησης των υποεξέταση θεμάτων. Και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν ε, είναι δικαιολογημένο αυτό, αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία τίθενται. Και επανερχόμεθα στο θέμα το οποίο συζητήσαμε σήμερα για τον έλεγχο μέσω της επικουρικότητας. Πολλοί δεν είναι πολύ σίγουροι γι' αυτό γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι το τεχνικό, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και μου άρεσε αυτό το οποίο είπε ο Χόρμπετ ότι το θέμα είναι η ουσία. Θα πρέπει δηλαδή να συζητήσουμε την πολιτική, να ασχοληθούμε ξανά με την πολιτική και βλέπουμε ότι όπου κινητοποιούνται τα κοινοβούλια, βλέπουμε ότι τα θέματα αυτά έχουν συγκεκριμένη σημασία. Βλέπουμε ας πούμε τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στα πλαίσια λοιπόν και του ελέγχου της επικουρικότητας υπάρχει μια κάποια κινητοποίηση για τα πολιτικά θέματα και όπως σας είπα πριν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικό μέτρων τα οποία φαίνονται μη πολιτικά και τεχνικά. Απαιτείται λοιπόν μια επανεισαγωγή της πολιτικής στη συζήτηση. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Τώρα, σε σχέση με την επικορικότητα, για σε ποιο βαθμό είναι πραγματικό πρόβλημα και το αν θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός κόκκινης κάρτας. Αν το δούμε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της διαδικασίας ε, έτσι όπως έχει προταθεί μέχρι τώρα, μερικές τροπολογίες ε, μπορεί να λειτουργήσουν θετικά. Το είδαμε ε, και φέτος ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας κατεπήγον τρόπος επιβράδυνσης κάποιων διαδικασιών. Όπως όταν είσαι πάνω σε ένα τραμ, δεν χρησιμοποιείς ποτέ το φρένο ασφαλείας. Έτσι λοιπόν και τώρα είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικά χρήσιμο, το οποίο πρέπει να συζητηθεί, αλλά μπορεί να έχει και αρνητικό συμβολικό χαρακτήρα γιατί για μια ακόμη φορά είναι ένα μέσο αρνητικό αντίθετα με άλλα μέσα τα οποία θεωρούνται επικοδομητικά όπως οι τροπολογίες. Για την διάδραση ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να συνεδριάζουν σε επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν έχω τα δεδομένα και για τα 28 κράτη-μέλη. Εδώ θα μπορούσαμε να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο οι πανεπιστημιακοί. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε όλες τις χώρες. Σε ορισμένα κοινοβούλια τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ιδιαίτερα περιορισμένο χρόνο ομιλίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο και είναι κάτι το οποίο θα καταστεί θα έλεγα κοινή πρακτική. Το πλεονέκτημα είναι ουσιαστικά ότι και τα μέσα ενημέρωσης θα ενδιαφερθούν για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο κοινοβουλίων. Ευχαριστώ επίσης και για την Ιταλική περίπτωση. Πράγματι είναι γενικού τύπου οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Υπάρχουν κάποιες πιο εξειδικευμένες μορφές συμμετοχής σε ορισμένες χώρες, όμως για μια ακόμη φορά σε περιπτώσεις όπως η Σουηδία και η Δανία γίνονται κάποιες συζητήσεις σε βάθος, σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν είναι κανόνας. Σχετικά τώρα με το πλεόνασμα πληροφόρησης. Όταν έκανα τη μελέτη για το Αυστριακό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια, πριν από τη Λισαβόνα, ένα από τα σχόλια τα οποία είχαν ακουστεί είναι ότι παίρνουμε τόσες πολλές πληροφορίες που πνιγόμαστε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο άπτεται της επιλογής των πληροφοριών και των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους τα εθνικά κοινοβούλια αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες αυτές και το μέγεθός τους την πληθώρα τους. Θα πρέπει σαν παράδειγμα να γίνεται ένας κατάλογος όλων των προτάσεων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπογραμμίζονται το πού, όχι σε δεσμευτικό επίπεδο, αλλά πού σε νομικό επίπεδο θα μπορούσαν να υπάρχουν θέματα ανησυχίας για την επικουρικότητα. Και εκεί να υπάρχει επεξεργασία. Για το θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ένα από τα βασικά πολιτικά θέματα αμφισβητεί κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται και κλεισμένων των θυρών, λόγω της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, λόγω της αυξημένης αποτελεσματικότητας, μόνο του ότι απαιτείται να λαμβάνονται αποφάσεις. Και από την άλλη υπάρχει το θέμα του υπολόγου, του ελέγχου, της ανάληψης ευθύνης. Και εδώ υπάρχει θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικό και είναι σημαντικό οι ακροάσεις αυτές να δείχνουν προς τα έξω το τι πραγματικά συμβαίνει και να βελτιώνουν και την κάλυψη των δεδομένων αυτών από πλευράς του τύπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ορισμένες αποφάσεις λαμβάνονται από τη μία. Το θέμα είναι γιατί λαμβάνονται και κλεισμένων των θυρών. Τα κοινοβούλια λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Καθηγητή Ροζεμπερκ, ευχαριστώ για τι ερωτήσει με τη σειρά. Θα απαντήσω γρήγορα. Σε σχέση με τον κύριο από την Τουρκία που ρώτησε για τη συμμετοχή στι εκλογέ. Εγώ θα το έβλεπα κάποιο πιο θετικά. Βάσει τη συμμετοχή στι ευρωπαϊκέ εκλογέ, Πρέπει να πούμε ότι διευρύνθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν και νέε χώρε μέλη, ε, με μεγαλύτερη αποχή για διάφορου λόγου στι εκλογέ. Δηλαδή αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που επιφέρουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αν εξαιρεθούν βλέπουμε ε, ε, ότι σε 35 χρόνια έχει μειωθεί κατά 10% που είναι αντίστοιχο αυτό ποσοστό με τις εθνικές εκλογές της χώρες αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλό θα ήταν να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για αυτό το θέμα. Βεβαίως δεν μπορεί να χαίρεται κανείς ε, όταν υπάρχει τόσο χαμηλή συμμετοχή, αλλά δεν είναι κάτι που αφορά ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις εθνικές εκλογές ε, από την οικονομική κρίση και μετά βλέπουμε να κυριαρχούν ευρωπαϊκά θέματα στις εθνικές εκλογές. Επιτέλους, στις κάτω χώρες, στη Σλοβακία, στη Γαλλία το 2012, στην Ιταλία σε όλες αυτές τις εκλογές που μπορεί να είναι βουλευτικές, ε, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά θέματα, συζητούν μεταξύ τους ε, στα debate ευρωπαϊκά θέματα οι υποψήφοι κτλ. Σε σχέση με τη συνάδελφα από τη Ρουμανία, που είπε ότι ήμασταν ε, αυστηροί, κακοί με τη Ρουμανία. Μπορεί, εμείς έχουμε στοιχεία μέχρι το τέλος του 2012 και ελέγχονται τα στοιχεία. σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στα ευρωπαϊκά θέματα, ποιο είναι το ζήτημα. Ε, θα πρέπει οι πολιτικές ελίτ να ασχολούνται με την Ευρώπη, να κάνουν κτήμα τους στα ευρωπαϊκά θέματα και να τα ε, λένε και στον τύπο όλα αυτά, στα μέσα ενημέρωση. Ο καθένας προβληματίζεται και αναρωτιέται τι γίνεται στη χώρα του, πέρα από τα στοιχεία και τις διαδικασίες. Ε, τι γίνεται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Γαλλία οι πολιτικοί ασχολούνται πραγματικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, έχουν επίγνωση, δρούν, ε, μια φορά τα επηρεάζουν, τα προωθούν, τα προβάλλουν και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Το δυστυχώς δεν είναι πάντα θεντικά. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ τώρα δυστυχώς αποχώρησε. Υποστηρίζει κάτι που ακούω σε επιχείρημα, μπορώ να σας πω ότι είναι κάπως κοινικό. Δηλαδή μπορούμε να δεχτούμε την κόκκινη κάρτα διότι το κατόφλι θα είναι τέτοιο ώστε δεν θα γίνεται χρήση μεγάλη συχνά ε, όπως έγινε και για τις κίτρινες κάρτες. Εντάξει, μπορεί να είναι ε, καλή διπλωματική λύση για να προσφέρουμε κάτι στον Κάμερον σε μια συζήτηση. Αυτό μένα με ενοχλεί λίγο. Γιατί είναι αυτή η στρατηγική του Τχομπλόγη, μπορεί να είναι και οφθαλμαπάτη. Ε, δηλαδή υποκρινόμαστε ότι δίνουμε εξουσία στα εθνικά κοινοβούλια, ενώ στην αλήθεια αυτό δεν ισχύει. Ε, η κυρία Όμεν ρώτησε για τις σχέσεις εθνικών κοινοβουλίων με τους ευρωβουλευτές. Η πρακτική διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι Γερμανοί ξέρουν πολύ καλά να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι του συμφέρει, γιατί είναι τόσοι πολλοί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του συμφέρει να συντονίζουν τη στρατηγική τους, γιατί ενδεχομένως μπορούν να ασκήσουν ε, πιέσεις και ε, είναι αρκετά ισχυρή η πολιτική και τα πολιτικά κόμματα στη Γερμανία ώστε να μπορούν έτσι να διασυνδέονται, να διακλαδώνονται. Στη Γαλλία, ας πούμε, είναι πιο ασθενή τα κόμματα. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι από τη Γαλλία. Από 577 βουλευτές, δύο είναι βουλευτές του Εθνικού Μετόπου, κάτω από 1%. Και θα ήταν δύσκολο να προσκαλούν κάθε φορά τους ευρωβουλευτές στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, γιατί η πρώτη ε, σε αριθμό κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευράς Γαλλίας είναι του Εθνικού Μετόπου σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κ. Ματιώτη, αν δεν απατάμε από την Ιταλία και συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Υπήρχε μια έλλειψη βαθιάς ανάλυσης, λέτε, των εθνικών κοινοβουλίων. Με πολύ πολιτικά ορθό τρόπο το διατυπώσετε. Δύο απαντήσει. Πρώτον, αυτό δεν ισχύει πάντα. Υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που έχουν ε, δημόσιες συνεδριάσει των επιτροπών του και μεταδίδονται και στην τηλεόραση τη και κάνουν πολύ βαθιά ε, ανάλυση. Δεν το γνωρίζουν πολύ αυτό, αλλά η Folketing ε, στη Δανία και κάθε Παρασκευή δείχνει τηλεόραση τις ε, επιτροπές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Αυτή η έλλειψη λοιπόν βαθιάς ανάλυσης που φαίνεται να επικρίνεται, επιτρέψτε μου λίγο να την υποστηρίξω. Είδαμε, με τεχνικό τρόπο μελετήσαμε ε, το πώς συζητούν τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, για την Τραπεζική Ένωση, ας πούμε, θα πρέπει να μπαίνουν στις τεχνικές λεπτομέρειες, το μέγεθος των τραπεζών, από ποιο επίπεδο και μετά ε, και ποιο μέγεθος τη σώζουμε ή όχι. Αλλά, ίσως δεν χρειάζεται να γίνεται και αυτή η συζήτηση, αλλά χρειάζεται και γενικότερη. Τι Ευρώπη θέλουμε, ε, μπορεί η Ευρώπη να γινεται και αυτη η συζητηση αλλα χρειαζεται και γενικοτερη τι ευρωπη θελουμε μπορει η ευρωπη να ελεγχει τις τράπεζες κτλ. για τον κύριο Χάουρεγγι για τις εντολές που δίνουν τα κοινοβούλες κυβερνήσεις. Νομικά υπάρχουν δύο χώρες η Δανία και η Αυστρία που δίνουν συγκεκριμένη εντολή στον Υπουργό και ο Υπουργό δεν μπορεί να το κουνήσει ούτε ρούπι. Η Αυστρία δεν το εφαρμόζει πάρα πολύ. Η Γερμανία θέλει να αλλάξει το σύστημα, μιλάει για εντολέ, αλλά προβλέπει και εξαιρέσει. Δηλαδή, η πιο σκληρή εντολή, α πούμε, υπάρχει μένα να είναι μόνο στη Δανία και μόνο για τι νομοθετικέ δραστηριότητε, όχι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχουν τέτοια εντολή με την νομική έννοια οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, γιατί δεν νομοθετούν. Προς το παρόν αυτό δεν έχει οδηγήσει σε εμπλοκές. Ακόμα και ο Φιλανδός Πρωθυπουργό, ας πούμε, δέχτηκε να βοηθήσει την Ελλάδα. Για τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ε, πώς να το πω, κάποια φορά εθνικά γυαλιά για να βλέπουν τα ευρωπαϊκά θέματα. Δεν ξέρω πώς δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Στο κάτω-κάτω αυτό είναι ο ρόλος του. Αν θέλουμε ευρωπαϊκή διάσταση υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το λόγο. Για ε, τις περιφερειακές βουλές που ρωτήσατε. Ναι. Στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης υπάρχουν ε, ε, σε πολλές χώρες, όχι μόνο σε ομοσπονδιακές χώρες, αλλά και στην Ισπανία και την Ιταλία υπάρχουν τοπικά κοινοβούλια που έχουν σημαντικές αρμοδιότητες για τον έλεγχο της επικουρικότητας και μπήκαν με πολύ ενθουσιασμό ε, σε αυτή την προσπάθεια σε πολλές χώρες γιατί επιτέλους τους ε, έδινε ιδιαίτερο ρόλο μια ευρωπαϊκή συνθήκη. Αλλά και αυτό γνωρίζει τα όρια του ως προς την επικουρικότητα και πώς ελέγχεται. σε τα όσα είπατε εσείς, ε, Υπουργέ. Είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών για τις πρακτικές τους μεταξύ των κοινοβουλίων. Γίνεται αυτό σε επίπεδο κόζακ. Αν υπάρχει κάτι που λειτουργεί σωστά ε, κοινοβουλευτικά στην Ευρώπη είναι αυτό. Και είναι λίγο κρίμα που η κόζακ ε, χρησιμοποιείται μόνο για αυτό σχεδόν και όχι για θέματα πολύ ίσως. Και επίσης με πολιτική ορθότητα διατυπώσατε ότι ε, τα εθνικά κοινοβούλια συνήθως ακολουθούν αυτά που αποφασίζουν οι ε, κυβερνήσεις. Μετά την οικονομική κρίση πολλές κυβερνήσεις έπεσαν μετά από προτάσεις δυσπιστίας, μορφής στο κοινοβούλιο τους και πολλές φορές ε, ε, έκτακτες. Όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά ζητήματα και οικονομικά υπάρχουν και κοινοβούλια που ρίχνουν κυβερνήσεις. Από την Ιρλανδία κάποιος ρώτησε, κύριος Χάνιγκαν, για την έκθεση των πέντε Προεδρών δεν γνωρίζω το θέμα επαρκώς για να το σχολιάσω. Για το δημοσιονομικό σύμφωνο, εγώ θα ήμουν κάπως πιο αισιόδοξο. Και ο συνάδελφος Φιλίππο Αργέ έδειξε μια αισιοδοξία. Σε πολλές χώρες ε, το δημοσιονομικό σύμφωνο και αντίστοιχες δομές είναι κάτι νέο. Ε, είναι εργαλεία που επιτρέπουν στα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν και στη Γαλλία και αλλού ε, ο πολιετής σχεδιασμός για τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι κάτι το καινοφανές. Βέβαια αυτό δεν είναι καμία τεράστια εξουσία στη Βουλή, αλλά γνωμοδοτούν, συζητούν καθόλου το εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο για ευρωπαϊκά θέματα. Και για τις ερωτήσεις της Πρόεδρου Χιούμπνερ για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα γιατί θέλουμε να είναι ανεξάρτητο αυτό το θεσμικό όργανο από τη φύση του αλλά και από κάπου ε, δεν πρέπει να ελέγχεται στη δημοκρατία. Εγώ εξεπλάγει και εκφράζω και δυσφορία ως Ευρωπαίος πολίτης. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα εθνικά για αυτό το θέμα. Το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου λέει ότι θα υπάρχει ένα φόρουμ που θα συνεδριάζει για τρεις φορές το χρόνο με εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και τώρα αυτό τίνει να καταντήσει μια πολύ σκοτεινή και τεχνική επιτροπή και είναι λυπηρό. Τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει αποκοινοτικοποιείται, δηλαδή ξεφεύγουμε από την κοινοτική μέθοδο και προχωρούμε προς τη διακυβερνητική. Αυτό είναι πρόβλημα μάλλον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Που δεν υπόκεινται σε αυτή την νομοθετική διαδικασία, αλλά είμαι βέβαιος ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια θα βρουν τρόπο να αντιδράσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και 25 χρόνια έχει μια παράδοση ανάληψης ευθυνών πριν του δοθούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες. Ε, αν δούμε πώς εξελίχθηκε η διαδικασία της συναπόφασης. Και είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά θα ε, καταφέρει να ελέγξει δημοκρατικά την Ευρωζώνη. Alors, pour la Για το θέμα των εκλογών Άκουσα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά πρέπει να επανατοποθετήσουμε το θέμα της αποχής σε μια ευρύτερη προοπτική τροποποίησης του δημοκρατικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά τις εθνικές εκλογές, αλλά και άλλες μορφές πολιτικής συμμετοχής. Παραπέμπω λοιπόν σε μια σειρά ερευνών που γίνονται εδώ και 30 χρόνια και δημοσιεύουν σε πενταετή βάση στοιχεία για τις δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρατηρείται εκεί ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση της συμμετοχής και της σχέσης με την πολιτική. Και οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν είναι παρά ένα στοιχείο από αυτήν την αλλαγή της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Δεύτερον, για το θέμα της επικουρικότητας. Ίσως να μην εκφράστηκα σωστά. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα στοιχεία βελτίωσης του ελέγχου της επικουρικότητας, αλλά στο περιεχόμενο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και εδώ, ίσως ήμουν βιαστικός πριν, αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις τεχνικές ελέγχου της επικουρικότητας. Θα πρέπει για τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταθούμε στο περιεχόμενο και στην ουσία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Αλλιώς να θυμίσω ότι δεν έχουν την ίδια αντίληψη τα εθνικά κοινοβούλια. Κάποια θέλουν να βελτιώσουν το σεβασμό αυτής της αρχής, βελτιώνοντας τη λειτουργία της Ένωσης. Άλλα κοινοβούλια έχουν άλλους στόχους. Θέλουν να μπλοκάρουν ίσως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θέλουν σε κάποιους τομείς να μπλοκάρουν κάποιες αποφάσεις. Για το θέμα της αποκοινοβουλευτοκοποίησης είναι ακαδημαϊκός ο όρος λίγο, αλλά θα συμφωνήσουν για τον ρόλο ακριβώς της απεξάρτησης, αν θέλετε. Τα κοινοβούλια, τα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν μέσα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν ή δεν ε, δεσμεύονται να τα χρησιμοποιήσουν. Έχουν πάρα πολλές δυσκολίες να τα χρησιμοποιήσουν τα μέτρα αυτά. Και αυτό είναι περίεργο. Να έχει κανείς μέσα στη διάθεσή του, αλλά να μην τα χρησιμοποιεί. Θα συμφωνήσω μαζί σας λοιπόν για την έννοια αυτή της απεξάρτησης, ορίμανσης ταυτόχρονα, αλλά ταυτόχρονα και μια τάση από κοινοβουλευτικοποίηση των διαδικασιών. Σχετικά τώρα με τις προτάσεις της εκθέσεως των Προέδρων. Ίσως εδώ κάποια σημεία να ενδιαφέρουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην έκθεση των Προέδρων η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο στόχος. Υπάρχουν πολλές παράγραφοι για τα Εθνικά Κοινοβούλια και υπάρχουν και κάποια και νέα σημεία. Παράδειγμα, απλό παράδειγμα το οποίο νομίζω θα μας οδηγήσει στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Προτείνεται να δημιουργηθεί μια συμβουλευτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συμπληρώνει και θα συντονίζει τα εθνικά συμβούλια τα οποία έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του Συμφώνου του Δημοσιονομικού. Γιατί το Συμβούλιο αυτό εφόσον υπάρξει γιατί να μην συνδέεται επίσημα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί σε αυτήν την μελλοντική πρόταση της Επιτροπής αυτής των Προέδρων να μην συνδεθεί λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί οι εθνικές δημοσιονομικές ε, επιτροπές να μην συνδέονται με τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί εδώ βλέπουμε ε, μια λειτουργία των κοινοβουλίων να έχουν στη διάθεσή τους μία θα έλεγα ποσότητα επαϊοσύνης έτσι ώστε να ελέγχουν πράγματα όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και στο ευρωπαϊκό. Να λοιπόν ένα σχόλιο για την πρόταση, την λεγόμενη πρόταση των Προέδρων. Αυτό μας οδηγεί στην Τραπεζική Ένωση, στην ανεξαρτησία, την αλληλοεξάρτηση κτλ. Εδώ έρχομαι σε αυτά τα οποία είπε ένας Βρετανός συνάδελφος αν θυμάμαι, γιατί να μην επισημοποιήσουμε περαιτέρω τις συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεκτικό Συνέδριο από τη μία, την Κεντρική Τράπεζα από την άλλη και τα Εθνικά Κοινοβούλια με τα αντίστοιχα όργανα σε εθνικό επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι συγγνώμη απλά σε συμφωνίες συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης, αλλά ε, στοιχεία ποσοτικά τα οποία θα επιτρέψουν για τα 3, 5, 6 επόμενα χρόνια μια τακτική αν θέλετε μορφή αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου σεβόμενη πάντα την ανεξαρτησία των συγκεκριμένων οργάνων. Στόχος της επισημοποίησης αυτών των συμφωνιών είναι η επανασύνδεση στα πλαίσια της αμοιβαίας βέβαια μορφή σεβασμού, αναγνώριση μάλλον των μεν από τους δε. Όλα αυτά περιλαμβάνονται και στην έκθεση του ΩΣΑ, δεν έχω χρόνο να την παρουσιάσω. Η οργάνωση αυτή στην έκθεση της ζητά να υπάρξουν τέτοιου είδους συμβάσεις, αν θέλετε, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα υπόλοιπα όργανα. Στην έκθεση του ΩΣΑ του 2014 περιλαμβάνεται επίσης κάτι άλλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί να μην δημιουργηθεί πέρα από την Κοζάκ ή μέσα στην Κοζάκ ένα μόνιμο μέσο συζήτησης των δημοσιονομικών πολιτικών. Μια υπηρεσία δηλαδή η οποία θα συγκεντρώνει και πληροφορίες αλλά δεν θα μένει σε αυτό. Είναι μια υπηρεσία η οποία θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη προς τα Εθνικά Κοινοβούλια και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέλος, για το θέμα της διακυβερνητικής μεθόδου από τη μία και της κοινοτικής από την άλλη. Μπορούμε να κατανοήσουμε τους όρους και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με κατεπήγοντα τρόπο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στα πλαίσια της διακυβερνητικής μεθόδου στα τελευταία σύμφωνα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Ταυτόχρονα τα εθνικά κοινοβούλια δεν ήταν ικανά να συνεισφέρουν ό,τι χρειαζόταν στα πλαίσια της διακυβερνητικής συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχασε λοιπόν διότι γίνονται όλα εκτός κοινότητας, αλλά τα εθνικά κοινοβούλια δεν κέρδισαν και τίποτα, εκτός αν πει κανείς ότι περιθωριακά και μόνο υπάρχουν ορισμένα θετικά στοιχεία. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση του ΟΣΑ του 2014. Λοιπόν για να επανέλθω τώρα σε αυτά τα οποία έλεγαν οι συνάδελφοι, πράγματι μπορεί να κρίνει κανείς την κατάσταση <clears throat> είτε λίγο θετική είτε λίγο αρνητική. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να εφεύρουμε. Υπάρχουν νέες μορφές σχέσεων ανάμεσα στα εθνικά και στα κοινοτικά όργανα. Και κυρίως πολιτικοποιώντας τις πολιτικές τις οποίες ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως στον οικονομικό τομέα θα μπορέσουμε να καλύψουμε την κρίση αντιπροσωπευτικότητας. Δεν θέλω να μιλήσω για δημοκρατικό έλλειμμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Μπρέσο. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο αγαπητός συνάδελφος. Δεν είπα ποτέ ότι είπατε κάτι άσχημο για τη Ρουμανία και τα λοιπά, ότι δεν είπατε την αλήθεια. Απλά σας ε, είπα ότι τα στοιχεία έχουν αλλάξει από το 2012, τώρα έχουμε 2015, υπάρχουν καινούργια στοιχεία και είπα μόνο ότι ήταν άδικο και το τονίζω αυτό άδικο να ασκήσετε κριτική στην Επιτροπή μου όταν η Επιτροπή μου είναι από τις πιο δραστήριες. Και όπως είπα επίσης, ε, εμείς κάθε μήνα κάνουμε δημόσια διαβούλευση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το μόνο μου σχόλιο ήταν αυτό. Εάν μας είχατε πει ότι η βάση δεδομένων στην οποία βασιστήκατε ήταν πρόσφατη, δεν θα το έκανα αυτό το σχόλιο. Αλλά αναφέρομαι, όχι τρία χρόνια πριν, αναφέρομαι στο τώρα. Και το είπα αυτό γιατί ε, μάλιστα εκφράσατε κάποια παράπονα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και χρειάζονται δύο χρόνια για να καταλήξουμε κάπου. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Είναι ενδιαφέρον να έχουμε συζήτηση πανεπιστημιακών με πολιτικούς ανάμεσα του στον ακαδημαϊκό και στον πολιτικό κόσμο. Ε, το ευχαριστιέμαι αυτό συζήτηση, αλλά υπάρχει μια διαφορά νοοτροπίας κουλτούρας. Εμείς ε, παρουσιάσαμε μια έρευνα που τελείωσε το 2011. Ως πανεπιστημιακή σημαίνει ε, ότι γρήγορα ε, συλλέγουμε και αναλύουμε στοιχεία. Κατανοώ ότι για την πολιτική ζωή χρειάζονται πιο ε, ενημερωμένα στοιχεία, πιο επίκαιρα, μάλλον κάποια διαφορά κουλτούρας είναι στη καινοτροπία. Ευχαριστώ. Έλμαρ, πριν κλείσουμε, μήπως θες να πεις τίποτα. Ναι, είμαι βέβαιη ότι είχες και άλλα να πεις και άλλες συναντήσεις και τα ναι, ευχαριστώ πολύ. Όντως, μόλις είχα στο γραφείο μου τον Πρωθυπουργό του Κωσόβου, καταλαβαίνετε, που έχει έρθει στις Βρυξέλλες σήμερα και είναι αρκετά δύσκολο και από πλευράς διεύρυνσης και από πλευράς μετανάστευσης ε, το θέμα αυτή τη στιγμή. I'm thankful that I had got a lot of... Ευχαριστώ πολύ. Συνέλεξα πολλά στοιχεία και ιδέες και από τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και από τους εμπειρογνώμονες. Myself. Ε, και η Mercedes, Μπρέσο και εγώ θα τα σημειώσουμε και θα τα συμπεριλάβουμε στις προτάσεις για την, στην γνωμοδότησή μας. Και η Γραμματεία θα μας δώσει και εκείνη διάφορες ιδέες. Γι' αυτό η Mercedes και εγώ ε, θελήσαμε να διευρύνουμε τη συζήτηση, όχι απλώς ε, να κάνουμε ένα σχέδιο έκθεσης, αλλά ένα έγγραφο εργασίας για να είναι πραγματικά μια βάση ε, και κυρίως γι' αυτό διεξήχθη η παρούσα ακρόαση. Και όταν μιλάμε για την πιο ισχυρή χρήση και αξιοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας, είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο για πρακτικούς λόγους και έχει σημασία να ακούγεται και η φωνή του Εθνικού Κοινοβουλίου κάθε φορά το εκάστοτε και να ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και τι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν έχει νόημα να κάνεις μεγαλόπνοες και φιλόδοξε προτάσεις όταν οι άλλοι είναι απέναντί σου ενωμένοι, μπλοκ, ένα μέτωπο. Δεν έχει νόημα αυτό. Ωραία. Πολλά ακούσαμε και θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσετε και το σχέδιο εκθεσής μας. Πρόεδρε αν συμφωνείτε, να το στείλουμε και στα Εθνικά Κοινοβούλια, το σχέδιο έκθεση, στου εμπειρογνώμονε. επίσης για να μας δώσουν την αίσθησή τους, τι απόψεις, τις τροπολογίες, ιδέες, ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι ώστε να επανέλθουμε. Να υπάρχει ένα feedback. Μέσα σε λίγες εβδομάδες να μας θέλετε και τις δικές σας προτάσεις να έχουμε την αίσθηση κάπου ότι είναι κοινό το εγχείρημα και η μοίρα. Ευχαριστώ πολύ Έλμαρ. Η γραμματεία σημειώνει και όχι μόνο. Ε, είναι και στο διαδίκτυο web stream η συνεδρίαση αυτή και μπορείτε να τρέξετε. Έλμαρ, τα σημεία 9 και 10 της έκθεσης ακούστηκαν πολλές φορές και θα πρέπει να δοθεί μάλλον ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους τρεις εξέχοντες εμπειρογνώμονες καθηγητές μας. Ε, εκτιμούμε πάρα πολύ το έργο σας και τις παρουσιάσεις σας. Ήταν πάρα πάρα πολύ χρήσιμες και χάρηκα πολύ που καταφέρατε να έρθετε εδώ στη σημερινή συνεδρία και συζήτηση με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα τα ξαναπούμε σε αυτό το διάλογο τον διακοινοβουλευτικό του χρόνου. Άπαξε της διεξάγεται αυτός. Αλλά δεν θα χαθούμε. Στο μεταξύ έχουμε και επισκέψεις 2-3 του χρόνου σε κράτη-μέλη ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και αν είστε διαθέσιμοι, διατεθειμένοι, ε, μπορούμε να έρθουμε να συνεδριάσουμε μαζί σας, στις επιτροπές σας, στα κοινοβούλια σας, εμείς με μεγάλη χαρά. Και αυτό που πρότεινε ο Έλμερ ήθελα να το πω κι εγώ όταν υπάρχουν σημαντικά ζητήματα να τα συζητούμε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, των εργαστηρίων ή των επιτροπών και να σας ενημερώνουμε. Γιατί καμιά φορά περνάτε και από τις Βρυξέλλες, σας φέρνει εδώ ο δρόμος σας και άτυπα και σε ατομικέ επισκέψεις ανεπίσημες θα είστε ευπρόσδεκτοι. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω κλείνοντας και να πω ότι ελπίζω να είναι ένα πρώτο βήμα σε μια μακρά συνεργασία για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και σημασίας και κυρίως για τους πολίτες. Γιατί αυξάνεται έτσι η δημοκρατική νομιμοποίηση όλων όσα αποφασίζονται και γίνονται παντού στην Ευρώπη. Και η συνεργασία μας είναι χρήσιμη και τεράστια σημασία πέραν της κανονικής καθημερινής δουλειάς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο θόρυβος, είναι η οθόνη που ανεβαίνει. Ε, μήπως είναι κανένα ξυπνητήρι για να τελειώσει η συνεδρία. Σε ευχαριστώ. Λύεται τη συνεδρία.